Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε στην ώρα μας. Καταρχήν έχουμε την έγκριση της ημερήσιας διάταξης αλλά έχω και μια μικρή τροποποίηση να σας προτείνω στην ημερήσια διάταξη. Ξέρετε ότι ότι ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι θα έρθει στις 9.30 να μας μιλήσει, περίπου στις 9.30 εν πάση περιπτώσει, και θα εξετάσουμε το budget review, το έγγραφο για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού και όλα τα συναφή θέματα. Γι' αυτό η πρότασή μου είναι να τροποποιήσουμε λιγάκι την ημέρηση διάταξη και συγκεκριμένα το σημείο 5 να το θέσουμε στη θέση του 3 ώστε ο Σαλβαδόρ μπορεί να, να μπορέσει να κάνει μια εισαγωγή στο έγγραφο αναλογισμού του, αναστοχασμού του μάλλον. ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα στη συνάντηση με τον κύριο Επίτροπο. Δηλαδή να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε το σημείο 3 και στην ε, επαφή μας με τον κύριο Επίτροπο. Χθες πάντως στην συνάντηση συνδιαλλαγής άκουσα ότι ορισμένοι συνάδελφοι θα θέλαν να αναφερθούν σε ορισμένα σημεία του πακέτου αναθεώρησης του προϋπολογισμού. Δεν τους βλέπω αλλά θα έρθουν κάποια στιγμή. Και έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε μαζί με τον κύριο Λεβαντόφσκι μια συζήτηση και για αυτές τις πτυχές. Συμφωνείτε λοιπόν <clears throat> να προτάξουμε το σημείο 5 στη θέση του σημείου 3. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Οπότε ούτως απεφασίστη. Ανακοίνωση της Προέδρου τώρα. Δεν έχω τίποτα να σας πω το ιδιαίτερο. βρισκόμαστε στο διαδίκτυο όπως ήθιστε. Δεύτερον, οι συντονιστές θα συντονίσουν Συγγνώμη. Οι συντονιστές έχουν εκπονήσει ένα σχέδιο εργασίας για το επόμενο έτος και αφού κλείσουμε την πρώτη φάση εργασίας μας με τα οριζόντια θέματα θα ασχοληθούμε με τα τομεακά θέματα, τα κατατομής θέματα. Θα αντιμετωπίσουμε τη γεωργία, την συνοχή και την αλληλεγγύη και μετά τις υπόλοιπες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατηγική Ευρώπης 20 στρατηγικές που υποστηρίζουν την, ε, το σχέδιο για την Ευρώπη του 2020 Και το ερώτημα βέβαια είναι μετά, είναι ακόμα λιγάκι επίμαχο, ποιες άλλες πολιτικές συμμετέχουν σε αυτή την προετοιμασία, έρευνα και καινοτομία, ε, διευρωπαϊκά δίκτυα κτλ. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε και για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, σχέση μας με τους πολίτες, ακόμα και με τα διηγητικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η δίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τύχει χρηματοδότηση. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε, όχι βέβαια σε μια πλήρη συνεδρία, ίσως, αλλά μία ώρα, τρία τέταρτα, πρέπει να αναφερθούμε και στα διοικητικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. <clears throat> Τρίτον, έχουμε μιλήσει ήδη για την ακρόαση. Νομίζω ότι έχετε όλοι στον φάκελό σας τα στοιχεία της ακρόασης αυτής. Δεν έχουμε ακόμα ονόματα. Αλλά ακόμα και αν σας είχαμε δώσει κάποια ονόματα χθες το βράδυ, μπορεί σήμερα να μην ήταν, να μην ήταν έγκυρα πια. Γι' αυτό περιοριστήκαμε να σας δώσουμε τη δομή της ε, ακρόασης. Η Γραμματεία έχει λάβει υπόψη τις προτάσεις όλων των πολιτικών ομάδων για την ακρόαση αυτή και ήταν πολλές αυτές τις προτάσεις. Και Έχουμε στείλει σε όλους προσκλήσεις για την ε, ακρόαση. Ορισμένοι είπαν «Ε, δεν θα μπορέσουν, άλλοι είπαν μπορούν. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τον οριστικό κατάλογο αυτών που θα είναι διαθέσιμοι να έρθουν στην ακρόαση και να συζητήσουν τα ζητήματα αυτά που μας ενδιαφέρουν. Τέταρτη ανακοίνωση και τελευταία. Συμφωνήσαμε με τους συντονιστές ότι θα κάνουμε μία γραμματολογική συζήτηση σε σχέση με τον τίτλο της εργασίας μας. Νομίζω ότι έχουμε όλοι εμπειρία από τέτοιες ενέργειες στη ζωή μας στο παρελθόν. Συμφωνήσαμε τελικά σε μια πρόταση που έκανε ο εισηγητής. Ο εισηγητής ζήτησε από όλες τις πολιτικές ομάδες να στείλουν τις προτάσεις τους και μετά θα τις κοιτάξει τις προτάσεις των πολιτικών ομάδων ο εισηγητής και θα κάνει μια πρόταση δικιά του μετά και θα μπορέσουμε στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών να συζητήσουμε περί του τίτλου. Εγώ θα ήθελα να έχουμε ένα σύντομο και πιασάδικο τίτλο. Γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω τον ε, κύριο εισηγητή να δεχθεί όλες τις προτάσεις των πολιτικών ομάδων και να τις συνθέσει σε ένα πάρα πολύ μακροσκελή τίτλο, αλλά να βρει κάτι το οποίο θα είναι πιο σύντομο. Αυτή λοιπόν ήταν η τελευταία μου, προτελευταία μου ανακοίνωση, τελευταία ανακοίνωση τώρα. Είπαμε πάντα ότι πρέπει να συνεργαστούμε και με τα Εθνικά Κοινοβούλια. μια πλήρη συνάντηση με τα εθνικά κοινοβούλια δεν πρόκειται να μας οδηγήσει πουθενά γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι μια σειρά από και δεν γίνεται ποτέ συζήτηση, δεν έχουμε ποτέ χρόνο να συζητήσουμε με τους ομολόγους μας από τα εθνικά κοινοβούλια. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι έτοιμοι να έρθουν στις Βρυξέλλες από τα Εθνικά Κοινοβούλια ή το Στρασβούργο, φυσικά θα τους υποδεχτούμε με μεγάλη χαρά. Έχουμε από την Πολωνική Σέμια ήδη ένα μεγάλο γκρουπ το οποίο ήρθε και έχουμε συζητήσει μαζί τους ποιες ήταν οι προθέσεις τους, ποιες ήταν οι προσδοκίες τους από, από εμάς και εμείς είπαμε τι περιμένουμε και εμείς από αυτούς μέσα στο δικό τους κράτος μέλος. Αλλά θα αποστείλω και μία επιστολή στις επιτροπές οι οποίες είναι αρμόδιες για τα ευρωπαϊκά θέματα στα εθνικά κοινοβούλια ώστε να τους προσκαλέσουμε και πάλι ακόμα και αν δεν μπορούν να έρθουν προσωπικά στις συνεδριάσεις μας, τουλάχιστον να μας αποστείλουν τις απόψεις τους. Και τις επόμενες μέρες θα αποστείλω αυτήν την επιστολή και επομένως απαντώ έτσι στο ερώτημα που διατύπωσαν ορισμένε συνάδελφοι. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ο James. Δύο πολύ σύντομα σχόλια για τα στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας που θα μελετήσουμε το κείμενο για το μήκος των δημοσιονομικών προοπτικών. Είναι σημαντικό για μας τους προπολογισμού, αλλά και για το Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα με βάση προτάσεις του Επιτρόπου Λεβαντόφσκη. Γιατί δεκαετής προοπτικές. Αυτό ούτε καν το σκεφτόμασταν στο Κοινοβούλιο. Είναι εντελώ αντίθετο με αυτό που είχαμε κατά νου θέματα ουσίας, νούμερα να το συζητάμε, αλλά να ξέρουμε και το, τη χρονική διάρκεια. Ίσως ο εισηγητής θα μπορούσε να μας κάνει ένα κείμενο προς μελέτη κάπως νωρίς, εφόσον είναι και της δικής του ευθύνη. Δεύτερον, για την ακρόαση. Μιλάμε για το Ένωση 2020 Καλό θα ήταν είχαμε και ορισμένε εξωτερικέ απόψει τι συμβαίνει η παγκόσμια διακυβέρνηση για το 2020. Έτσι ώστε να μην βρεθούμε σε ένα σκηνικό που θα έχει αλλάξει εντελώ η φύση του πέριξ περιβάλλοντο τη Ένωση. Αυτοί που δουλεύουν για τις μακρόπνες τάσεις, χθε είχαμε στην Επιτροπή Εξωτερικών, είχαμε ένα θέμα για την διακυβέρνηση με βάση το 2020. Ναι, πράγματι υπήρξαν πολλές προτάσεις σχετικά. Νομίζω ότι η γραμματεία μας προσπαθεί στο βαθμό του δυνατού να τις συνθέσει με τον πιο ισορροπημένο τρόπο και να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό εγκάρσια. Αλλά βέβαια πρέπει ό,τι προτάσεις έχετε να μας τις διαβιβάσετε. Σε ό,τι αφορά τώρα το μήκος. Έχουμε ήδη συζητήσει για το σχέδιο δράσης για το 2011 πριν από δύο εβδομάδες και είπαμε ότι το Δεκέμβριο στις 6 Δεκεμβρίου θα συζητήσουμε για τα θέματα του μήκους των δημοσιονομικών προοπτικών, της διάρκειας μάλλον τους. Θα έρθει ο Σαλβαδόρ λοιπόν με τον ποναμά του Αγίου Νικολάου και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ερχόμαστε στο σημείο 5, το οποίο πια είναι το σημείο 3. Έχουμε όλοι στα χέρια μας το νέο έγγραφο αναστοχασμού το οποίο μας έχει παρουσιάσει ο Σαλβαδόρ Γκαρίγα. Νομίζω ότι το έχετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, αν δεν το έχετε ήδη εντύπωση και θα δώσω το λόγο κατευθείαν στο Σαλβαδόρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μερικές ε, σύντομες σκέψεις για τον τίτλο όπως ε, είπατε εσείς. Η άποψη του εισηγητή ήταν να είναι το δυνατότερο σύντομος ο τίτλος της έκθεσης που θα προέλθει από την Επιτροπή μας, αλλά τελικά πρέπει να είναι <clears throat> συνενετικός αυτός ο τίτλος μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων και το μόνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι θα ξεπεράσει τις τρεις αράδες ο, ο τίτλος. Αυτός καταλαβαίνετε τώρα πόσες λέξεις μπορεί να περιέχει ο τίτλος. Εγώ θα ήθελα μια απλή φράση και θα έφτανε αυτό. Το έγγραφο τώρα το που σας παρουσιάζω έχει μερικά πιο τεχνικά χαρακτηριστικά και έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εξελιχθεί ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης συνδιαλλαγής ανέφερε ο πρόεδρος Λαμασούρ της Επιτροπής Προϋπολογισμών ότι το σύνολο των κονδυλίων που δεν εκταμιεύθηκαν και γύρισαν στα κράτη-μέλη έφτασαν τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια. Πάνω από το 1 τρίτο ενός ετήσιου προϋπολογισμού λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι τα θέματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξακολουθούν να είναι επίκαιρα και σημαντικά. Γιατί εξακολουθούμε να αφήνουμε ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού χωρίς ικανοποιητική εκταμίευση. Και αυτό φυσικά έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Γιατί ήδη το άρθρο 317 της ε, Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτελεί τον προϋπολογισμό και με συμφωνία των κρατών μελών, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Ένας προϋπολογισμός ο οποίος εν μέρη δεν εκτελείται και επανέρχεται, επανέρχονται τα κονδύλια στα κρατημέλη, δεν είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος καλύπτει ούτε από δημοσιονομική ούτε από πολιτική έποψη τους στόχους που έχουμε θέσει όπως αναφέρεται και στο οικείο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επειδή λοιπόν αυτό είναι μία από τις θεμελιώδεις πτυχές του προπολογισμού που έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε επίπεδο Επιτροπής Προπολογισμού και με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού έναντι της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η Επιτροπή ΣΟΥΡΕ. Εγώ τώρα θα ήθελα να ευχαριστήσω σε σχέση με το έγγραφο σκέψης τον ρόλο της γραμματείας. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα στον τομέα που αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών. Περιμένουμε ακόμα μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί. Ελπίζουμε ότι θα δοθεί στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το Νοέμβριο, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες λένε <clears throat> ότι στις αρχές Δεκεμβρίου και μόνο θα έχουμε αυτό το έγγραφο. γιατί αυτό είναι το έγγραφο στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της για απλοποίηση και οι οποίες φυσικά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο έγγραφο αναστοχασμού της Επιτροπής μας. Το έγγραφο αυτό θα αντιμετωπίσει και την σωστή διαχείριση και την ποιότητα των δαπανών και φυσικά θα πρέπει να προσθέσουμε καιρό και ορισμένα στοιχεία για την απλοποίηση, τη διοικητική απλοποίηση σε ό,τι αφορά την χρηστή διοίκηση και τον έλεγχο των δημοσιονομικών δαπανών. Στις σελίδες 2 και 3 έχετε τις βασικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να πριτανεύουν στην εκτέλεση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, την αποτελεσματικότητα, την ε, οικονομία, όλα αυτά είναι στοιχεία, την εξοικονόμηση είναι όλα αυτά στοιχεία τα οποία τονίζει και το ελεκτικό συνέδριο, όπως φάνηκε και στην πρόσφατη ακρόαση που διοργανώσαμε και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Υπάρχουν τρεις <clears throat> δυνατότητες οι οποίες προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, η συγκεντρωτική διαχείριση, η διαμεμοιρασμένη διαχείριση και η κοινή διαχείριση. Σε ό,τι αφορά την πρώτη, την συγκεντρωτική διαχείριση, από την πλευρά της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται αυτή η διαχείριση φυσικά και αφορά μια σειρά από κοινοτικού φορείς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Οι φορείς λοιπόν αυτοί <clears throat> έχουν βάσει αυτής της διαδικασίας τη δυνατότητα να αυτοδιαχειρίζονται και η διαχείρισή τους στη συνέχεια την χάνει ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο δεν επηρεάζει αυτή η διαδικασία. Πάντως αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό για την Επιτροπή μας, την ΣΟΥΡΕ, που είναι η λεγόμενη κοινή διαχείριση. Η κοινή διαχείριση, η, η καταμερισμένη διαχείριση καλύτερα, είναι αυτή η οποία καλύπτει περίπου τα 80% όλων των πολιτικών και όλων των δαπανών. Είναι πολύπλοκη αυτή η διαδικασία γιατί εκχωρείται η διαχείριση και το κομμάτι το, της εκτέλεσης του προπολογισμού στα κράτη-μέλη, τα οποία θα πρέπει να εκτελέσουν τις αντίστοιχες αυτές γραμμές του προπολογισμού και φυσικά αυτό συνοδεύεται από μια στενή παρακολούθηση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν την ευθύνη της διαχείρισης των κοινωτικών πόρων, εξασφαλίζοντας ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για ολοκληρωμένη διαχείριση και έλεγχο και ώστε να μπορέσει να υπάρξει το λεγόμενο DASI, λεγόμενη δήλωση αξιοπιστίας, θετική δήλωση αξιοπιστίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διεκδικήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια την ε, αναγκαιότητα της ε, θετικής δήλωσης αξιοπιστίας DAS. Αυτό όμως δεν γίνεται δυνατό ακόμα γιατί υπάρχουν προβλήματα με τους τελικούς αποδέκτες. Η καταμερισμένη λοιπόν διαχείριση συγκεντρώνεται περισσότερο αυτή τη στιγμή στην αγροτική πολιτική και την πολιτική συνοχή. Η πολιτική συνοχή που καλύπτει το 31% του ευρωπαϊκού πολιτισμού εξακολουθεί να είναι η πολιτική η οποία θέτει τα πιο σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και ιδίως προβλήματα σε σχέση με τον έλεγχο ο οποίος θα πρέπει να γίνεται από το ελεγκτικό συνέδριο. Παραμένουν σφάλματα και ελλείψεις στο, στην εκτέλεση του προϋπολογισμού που πολλές φορές δίνουν ελαβή και σε κριτική εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μέλων. Στην περίπτωση της Γεωργίας είναι πιο αποτελεσματικό το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης και ελέγχου και αυτό έχει οδηγήσει σε μια σημαντική ε, μείωση των ε, σφαλμάτων τα οποία έχουν ε, διαπιστωθεί από το ελεκτικό συνέδριο. Επομένω, οι εναλλακτικέ ε, προτάσει που εφαρμόσαμε στον αγροτικό τομέα έχουν λειτουργήσει πολύ καλά για να υπάρχει καλύτερη διαχείριση, καλύτερο έλεγχο των ε, διαρθρωτικών πόρων και των πόρων συνοχή. Χρειάζεται παρόλα αυτά να υπάρξει και πιο ε, έντονη δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συνεχιστεί η βελτίωση η οποία ήταν σημαντική τα τελευταία χρόνια. Και τέλος έχουμε τη λεγόμενη κοινή διαχείριση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με διεθνείς φορείς, <clears throat> όπως παραγωγός χάρη με συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, όπου και πάλι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Διακόπτεται ο μιλητής. Μας έχουν ε, δώσει στοιχεία τα οποία οδήγησαν σε τροπολογίες στο δημοσιονομικό μας κανονισμό για να υπάρχει καλύτερος έλεγχος των κονδυλίων που δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνείς οργανισμούς και των οποίων πολλές φορές τα ίχνη χάνονται. Δεν ξέρουμε λοιπόν κατά πόσο έχουν δαπανηθεί σωστά. Ε, έχουμε εμπιστοσύνη σε αξιόπιστους φορείς όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει σωστή διαχείριση όλων των κοινωτικών πόρων. Ένα πρόσθετο στοιχείο αυτής της από κοινού διαχείρισης είναι η έλλειψη ορατότητας των κοινωτικών πόρων οι οποίοι δίδονται μέσω τρίτων φορέων όπως είναι ο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερο χορηγός και σε όλους σχεδόν τους διεθνού οργανισμού. και παρόλα αυτά δεν φαίνεται ότι προέρχονται τα κονδύλια αυτά από την ευρωπαϊκή ορατότητα. Η ορατότητά μας είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μεγάλη σημασία όταν εμείς σκεφτόμαστε για το πώς θα προετοιμάσουμε τις επόμενες δημοσιονομικές όπως είπαμε και σε σχέση με το θέμα της ε, απλοποίησης, το οποίο θα πρέπει να προσθεθεί μεταγενέστερα στο έγγραφο αυτό όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε την ανακοίνωσή της. Ο στόχος μας δεν είναι μονάχα να εξασφαλίσουμε τη σωστή διαχείριση για να χρηματοδοτηθούν προγράμματα τα οποία δίνουν προσθέμενη αξία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εθνικές κοινέ γνώμες των κρατών μελών είναι αρκετά ευαίσθητες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ευρωπαϊκό προπολογισμό και ω εκ τούτου θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση του προπολογισμού και επίπεδο σφαλμάτων και ατασταλιών το οποίο να προσεγγίζει το μηδέν. Όταν είναι όλο και πιο δύσκολη η χρηματοδότηση, όταν έχουμε όλο και μεγαλύτερε εντάσει στα θέματα του προπολογισμού, είναι φανερό ότι η βελτίωση στην εκτέλεση και τον έλεγχο του προπολογισμού θα μα δώσει μεγαλύτερη ισχύ και επίσης θα μας δώσει και τη δυνατότητα να εξοικονομήσουμε περισσότερα κονδύλια του προϋπολογισμού αν αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα. Και φυσικά και το θέμα της αυλοποίησης επέχει μεγάλη σημασία. Όλοι σας είσαστε βουλευτές που έρχεστε από ευρωπαϊκές περιοχές και περιφέρειες που χρησιμοποιούν πόρους από τον προϋπολογισμό και οποιοδήποτε έχει σταθεί σε επαφή με κοινωτικά προγράμματα και κοινωνικά κονδύλια. Πάντα διατυπώνει το παράπονο αυτό ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις και οι κατευθυντήριες οδηγίες για κάθε πρόγραμμα, οι οποίες ποικίλουν από το ένα πρόγραμμα στο άλλο και είναι σε βάρος της ε, διαφάνειας και της αφήνειας των προγραμμάτων αυτών και μπορούν να οδηγήσουν σε σφάλματα. Πολλέ φορέ για διαφορετικά προγράμματα κοινοτικού χαρακτήρα υπάρχουν διαφορετικοί εκτελεστικοί κανόνε, κάτι το οποίο κάνει πολύ δύσκολο και τον εκτελεστικό έλεγχο και τον έλεγχο από την πλευρά, τον έλεγχο των μικρών αποδεκτών, <clears throat> των τελικών αποδεκτών, ιδίως όταν πρόκειται για, μεγάλου, για μικρούς δήμους και κοινότητες που δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν ενδελεχώς όλα αυτά τα στοιχεία. Επομένως, η Κομισιόν έχει την πρόθεση να προχωρήσει σε μια ευρεία διαδικασία απλοποίησης των κανόνων εφαρμογής αυτών των κοινοτικών προγραμμάτων με στόχο να μπορούν να ερμηνεύονται αυτοί οι κανόνες ε, εφαρμογής από τα κράτη-μέλη και να μην χρειάζεται να ζητά κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κανόνες ε, διαχείρισης και κανόνων και ελέγχου συγγνώμη, που είναι ανεδαφικοί. Πιστεύω ότι αυτή θα πρέπει να είναι η, οδηγή, η οδηγός γραμμή που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, η πολυπλοκότητα στη διαχείριση των κοινωτικών κονδυλίων δεν έχει μειωθεί, αλλά με την πάροδο του χρόνου έχει αυξηθεί. Πολλές φορές τα κοινωτικά προγράμματα δεν εκτελούνται γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τελικοί αποδέκτες οι οποίοι δεν θέλουν να διαδέξουν τον κίνδυνο να ζητήσουν κοινοτική χρηματοδότηση γνωρίζοντας ότι είναι τεράστια η πιθανότητα να, κάνουν, να υπάρξουν σφάλματα και να έχουν μετά νομικά προβλήματα με τη, τα κράτη-μέλη την Κομισιόν που διαχειρίζονται τα προγράμματα αυτά και προτιμούν να μην πάρουν τη χρηματοδότηση καθόλου. Τέλος, σε ό,τι αφορά την ποιότητα της εφαρμογής, οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, Βλέπετε στη σελίδα 6 μια σειρά από θέματα τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο σκέψης και ανοστοχασμού από τη δική μας πλευρά. Μέσα στη συζήτηση που ξεκινάμε σήμερα και θα ακολουθήσει και στις επόμενες εβδομάδες είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά την ποιότητα η απλοποίηση και η ενίσχυση των ε, εργαλείων εφαρμογής του προϋπολογισμού και αυτό θα πρέπει να γίνεται και ανάλογα με τις διάφορες πολιτικές και να εξασφαλίσουμε λοιπόν και ποσοτικοποιήσιμους στόχους και προστιθέμενη αξία. Η απροποίηση λοιπόν αυτή δεν θα μειώσει μόνο του, το, την πιθανότητα ασφάλματος, αλλά θα μειώσει επίσης και το συνολικό κόστος και χρειάζεται να έχουμε καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στο κόστος του ελέγχου και την αποτελεσματικότητα δηλαδή να έχουμε μια ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των ε, ελέγχων και ακόμα περισσότερο χρειάζεται μια βελτίωση στο μέλλον στις διαδικασίες <clears throat> διαχείρισης και παρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σας λέω και πάλι ότι αυτό είναι απλώς ένα εισαγωγικό έγγραφο κύριε Πρόεδρε. Ελπίζουμε <clears throat> ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να μας παράσχει ένα πιο ευρύ έγγραφο σε ό,τι <clears throat> αφορά τα θέματα της απλοποίησης και της βελτίωσης των διαδικασιών του προπορισμού που θα το λάβουμε στη συνεχεία απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Σαλβαδόρ. Απλώς ήθελα να σας υπενθυμίσω. Έχουμε δύο ακόμα θέματα, δύο ακόμα ε, συγγνώμη, έγγραφα με τα οποία θα πρέπει να ε, εργαστούμε, να τα εξετάσουμε <clears throat> την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που αφορά τη βελτίωση της ε, δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε επίσης από το Τμήμα Πολιτικών Μελετών ένα έγγραφο, μια ανασκόπηση κατά κάποιο τρόπο της κατάστασης των δημοσιονομικών προοπτικών και της εφαρμογής αυτών των ιδίων. <clears throat> και φυσικά δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση το έγγραφο αυτό στην ευελιξία με την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Βλέπετε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή όπως και στο παρελθόν υπήρξε στις δημοσιονομικές προοπτικές. Λοιπόν, ποιος θα ήθελε να λάβει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να θέσω τρεις ερωτήσεις προς τον αξιότιμο εισηγητή. Αν κοιτάξει κανείς τα τεχνικά παραρτήματα στις σελίδες 7 και 8 και αν προσπαθήσει να υπολογίζει, όχι απλά να δει δηλαδή, αλλά να υπολογίσει κανείς πώς έχουν τα πράγματα, θα δει ότι το ποσοστό εφαρμογής στη συγκεκριμένη περίοδο 7-8-9 είναι 2,5% χαμηλότερο από ό,τι στις, δημοσιονομικές, στις προηγούμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Μιλάμε δηλαδή για ποσοστό εφαρμογής απορρόφησης 96 ε, με 97, ενώ στην προηγούμενη περίοδο ήταν 98 και. Καλό είναι αυτό ή κακό, αυτό είναι το ερώτημα. <clears throat> Αν δεν έχουμε απάντηση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε αυτά προσεκτικά. Αν δει κανεί τι έγινε τα τρία πρώτα χρόνια των προηγούμενων δημοσιονομικών προοπτικών ξεκίνησαν από 85,89%. Ουσιαστικά λοιπόν τώρα είμαστε πιο χαμηλά αν το συγκρίνουμε με την πρώτη περίοδο των προηγούμενων δημοσιονομικών. Και επίσης αυτό το οποίο μπορεί να δει στη σελίδα 8 βλέπει ποιες είναι οι γραμμές όπου το ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο. Υπάρχουν τρεις τίτλοι. Το 3, 4 και 5. Έχουν απορροφηθεί πολύ χαμηλότερα, ε, πολύ λιγότερο από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι δύσκολο να εξηγηθεί αυτό το φαινόμενο. Και τέλος, σχετικά με τα λάθη που έχουν γίνει ή με τα ταμεία συνοχής. Η κατάσταση, ή μάλλον αυτό που μας αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό το οποίο εξετάζουμε δεν είναι το τι γίνεται τώρα. Το θέμα είναι να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι ακριβώς λογιστικές μελέτες έχουν γίνει και στόχος είναι να μειώσουμε τον αριθμό των λαθών, αλλά να μειώσουμε ταυτόχρονα και τον χρόνο εφαρμογής από 1,2 έτη σε 1,1 έτος. Θα ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή του εισηγητή στα δύο αυτά θέματα. Το θέμα είναι να αναλύσουμε τα παρατήματα, τα τεχνικά και να δούμε ότι τελικά αυτές οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν με την προηγούμενη περίοδο σε τι οφείλονται. Θα μαζέψουμε τα ερωτήματα πρωτού απαντήσει ο κύριος εισηγητής. Κύριε Καρβάλιου. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε την έκθεση της Ήτρε για την απλούστευση στα προγράμματα Έρευνα και καινοτομία ήμουν Γήτρια. Η έκθεση ψηφίστηκε στην Ήτρα. Όλε οι ομάδε την υποστήριξαν και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια στι Βρυξέλλε στι 11 Νοεμβρίου. Η Κομισιόν θα κάνει την απλούστευση αυτή σαν ένα είδος τεστ πριν επεκτείνει την μέθοδο αυτή απλούστευσης και σε άλλα προγράμματα. και μελετήθηκε το πρόγραμμα από την αρχή του. Από την αρχή που ορίζονται προτεραιότητες, επιλογή, έλεγχος, συμμετοχή των κρατών μελών στην έγκριση, ο πλήρης κύκλος. Και η ερμηνεία των κανόνων από τις διάφορες υπηρεσίες μέσα στην ίδια γενική διεύθυνση ή μεταξύ των γενικών διευθύνσεων διαφέρει η ερμηνεία. Χρειάζεται πολλή δουλειά λοιπόν για να είναι πιο προσβάσιμα τα προγράμματα. Η έκθεση είναι η αρχή μόνο. Το σημαντικό θα είναι η εφαρμογή εκ μέρους της Κομισιόν. Δύσκολο έργο. Αν όμως πετύχει αυτό το εγχείρημα στην Κομισιόν, Μερικές από αυτές τις ε, απλουστεύσεις, οι απλοποιήσεις καλύτερα, θα μπορούσαν να επεκταθούν ή να προσαρμοστούν και για τα διαρθρωτικά ταμεία. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σκέψεις και μία ερώτηση. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας δίνει ο εισηγητής και καλό θα είναι να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Δύο σημεία. Πρώτον, πάντα γίνεται μια τεράστια συζήτηση για τις διαφορές ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις πληρωμές. Γιατί συμβαίνει αυτό. Θεωρητικά ακαδημαϊκά, κανονικά θα έπρεπε ότι αποφασίζουμε να είναι 100% η εφαρμογή, χωρίς θεωρητικά, χωρίς καμία εξαίρεση. Αυτό θα έπρεπε ε, να γίνει στην καλύτερη των περιπτώσεων. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να δούμε γιατί δεν συμβαίνει αυτό. Βλέπω εδώ ότι ο εισηγητής ζητάει να αξιολογήσει την κατάσταση συνολικά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει η αξιολόγηση, να προσπαθήσουμε να ανοιχνεύσουμε τους λόγους γιατί οι υποχρεώσεις είναι χαμηλότερες από το σύνολο του προϋπολογισμού και οι πληρωμές ακόμα πιο χαμηλές και αυτό μάλιστα κρατάει χρονικά. Απαιτείται μια ανάλυση αυτού του φαινομένου γιατί διαπιστώνεται πάντα σε κάθε δημοσιονομικό έτος. Προσπαθούμε να φέρουμε τις πληρωμές ε, κοντά στις υποχρεώσεις. Εν μέρη μόνο πετύχαμε, αλλά ε, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και θα θέλαμε να έχουμε μια καλύτερη ανάλυση αυτού του προβλήματος. Μόνο αν υπάρξει πλήρης απορρόφηση τότε θα έχουμε ένα πλήρη έλεγχο ακριβώς των προοπτικών. Θα πρέπει όμως να έχουμε τη δυνατότητα αποκατάστασης των προοπτικών και σε σχέση με τα αποτελέσματα της προσπάθειας την οποία κάνουμε. Για το κοινωνικό ταμείο πρόσφατα υπήρξε ένας δημοσιονομικός ελεγκτής ο οποίος έκανε μια έρευνα σε βάθος σε όλες τις λεπτομέρειες αλλά τα αποτελέσματα τελικά αυτής της προσπάθειας δεν έγιναν γνωστά. Κανένας δεν έθεσε ερωτήματα γι' αυτό. Σαν παράδειγμα, το αποτέλεσμα ποιο θα ήταν για κάποιες πιστώσεις, να βάλουν τους μετανάστες στην αγορά εργασίας. Το πέτυχαν αυτό. Κανένας δεν ρώτησε αν ο στόχος επετέφθη. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει για να γίνει να υπάρξει μια πιο σωστή ανάλυση. Δεύτερον, ο κύκλος εφαρμογής. Και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε και αυτό έχει σχέση με αυτά που είπε ο Έλλης η διάρκεια του ΕΜΕΦ. Όταν έχουμε μία περίοδο για τα διαφορετικά ταμεία, ξέρουμε ότι τον πρώτο χρόνο δεν συμβαίνει σχεδόν τίποτα. Όλοι ασχολούνται με τον προγραμματισμό, τη σχεδίαση, την προπαρασκευή της γραφειοκρατίας κτλ. Το δεύτερο χρόνο κάπως αρχίζουν λίγο τα πράγματα να ανεβαίνουν. Τον τρίτο χρόνο ελπίζουμε να δουλεύει σχετικά καλά και τον τέταρτο χρόνο τα πράγματα να τρέχουν με όλη την ταχύτητα. Ε, ναι, αλλά αυτό είναι προβληματικό όμως. Αν πήγαιναν έτσι τα πράγματα τότε τον 7ο χρόνο θα έπρεπε ε, να τρέχουν τα πράγματα με τρομερή ταχύτητα και θα πρέπει ξαφνικά να τα διακόψουμε όλα και να ξαναρχίσουμε εκ νέου με το νέο κύκλο και να περιμένουμε πάλι κάποια χρόνια για να φτάσουμε σε μια ταχύτητα κρουαζιέρας λοιπόν. Αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός ο κύκλος, τι ακριβώς συμβαίνει τον πρώτο και τον δεύτερο χρόνο δεν είναι αποτελεσματικό δυστυχώς το σύστημα που χρησιμοποιούμε. Δεν είναι σωστός αυτός ο τρόπος των πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε κάτι να κάνουμε ακριβώς για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Επικαλυπτόμενες περίοδοι σαν παράδειγμα ή καλύτερη σε βάθος ανάλυση. Γιατί φοβάμαι ότι χρησιμοποιούμε στρεβλά πολλά από τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα διαρθρωτικά και σε άλλα ταμεία. Μπορούμε να βλέπουμε όχι μόνο τους αριθμούς των κύκλων εφαρμογής, αλλά να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Να δούμε αν θα πρέπει η επόμενη περίοδος εφαρμογής να είναι 5, 7, 10 χρόνια. Αν είναι να χάνουμε ένα, 2, 3 χρόνια για τη νέα προγραμματική περίοδο, δεν έχει νόημα να μιλάμε για 5 χρόνια ή για 7 μόνο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ανάλυση του κύκλου εφαρμογής πρώτα και μετά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μα είπε ότι θα ήσουν σύντομο. Αυτό δεν το έκανε όμως. Δεν τήρησε την υπόσχεσή σου. Θέλω να χαιρετήσω λοιπόν τον κύριο Επίτροπο. Καλώ ήλθατε κύριε Επίτροπε. Αλλά έχουμε ακόμα μερικού ομιλητέ ε, στον κατάλογο για τα υπόλοιπα θέματα. Λοιπόν, πάλι τονίζω, ο Ράιμερ θα μιλήσει πάρα πολύ σύντομα, όχι σαν τον Γέρον. Αυτή τη φορά θα μιλήσω πραγματικά σύντομα, γιατί έχουν ελεγχθεί πολλά από αυτά που ήθελα να καλύψω. Νομίζω ότι το ερώτημα της ε, ενδιάμεσης ε, αξιολόγησης των ε, προγραμμάτων και το θέμα της επικάλυψης στο χρόνο θα πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Θα έχουμε τις νέες ναυαρχίδες για την Ευρώπη του 2020, αλλά δεν πρέπει να τις υπερφορτώσουμε με έρμα από προηγούμενα προγράμματα. Και γι' αυτό ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε μαζί με τον εισηγητή αν για αυτό το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Κομισιόν μία σειρά από θέματα τα οποία έχουμε θέσει εμείς και να τα θέσουμε σαν απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτού αποδηθεί και σε νέες ασκήσεις φαντασίας και δημιουργικότητας η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ο Αλεξάνδρ Άλβαρο, πολύ όμως σύντομα, πολύ σύντομα. Βεβαίως κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ ευχαριστώ. Μετά από αυτά που είπε ο Γιώραν Φέρμ, εγώ συμφωνώ, το είπε και ο Ράιμερ, ώστε θα πρέπει να ελέγχουμε τους πόρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε κάθε φάση του κύκλου εφαρμογής. Αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνεπείς και με τον εαυτό μας. <clears throat> Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό μονάχα στη δική μας επιτροπή, όταν στη συνέχεια, όταν είμαστε επιτροπή προϋπολογισμού, θα πρέπει να ακολουθούμε μια αντίστοιχη αντιμετώπιση. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει και μια ένα έλεγχο αποδοτικότητα, όπω και ζητήσε ο Τζέμ Σέλ, παραδείγματο χάρη για του μη κυβερνητικού οργανισμού. Αυτό το είχαν απορρίψει. Το είχαμε απορρίψει στην Επιτροπή Προπολογισμών. Λοιπόν, αν υπάρχει ένα εκατομμύριο, ένα δισεκατομμύριο παραδείγματο χάρη το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για μη κυβερνητικού οργανισμού, όπω είπε ο Τζέμ Σέλ, τι θα γίνουν αυτά τα ποσά, πώ θα χρησιμοποιηθούν για άλλε δραστηριότητε, Λοιπόν, ό,τι λέμε εδώ θα πρέπει να είναι συνεκτικό και συνεπέ με αυτό που γίνεται στην Ολομέλεια και σε άλλε επιτροπέ. Ο Τζέμ, Έλες, ναι, θα λάβει το λόγο, αλλά έχω ακόμα τους υπόλοιπους ομιλητές που δεν τους έχουμε εξαντλήσει. Ο Έντι Γιάνν και μετά ο Τζέμ Έλες. Θα είμαι σύντομος κι εγώ. Καταρχάς νομίζω ότι συνδέεται το θέμα του αριθμού των κρατών μελών που ωφελούνται από κάποιες συγκεκριμένες γραμμές και τα θέματα ελέγχου. η συζήτηση που είχαμε είναι όλα τα ταμεία θα πάνε σε όλα τα κράτη-μέλη ή θα περιοριστούν σε κάποια κράτη-μέλη, ίσως εκεί θα μπορούσαμε να κερδίσουμε σε αποτελεσματικότητα. Σχετικά ε, με τον έλεγχο των αποτελεσμάτων και όχι μόνο των στοιχείων ε, τα οποία προηγούνται της εξέλιξης ενός προγράμματος. Σίγουρα και εδώ υπάρχει κέρδος σε επίπεδο αποτελεσματικότητα. Θυμίζω ότι η διεθνής διαφάνεια ε, έχει δημοσιεύσει ε, το, θα έλεγα, τον κατάλογο με τη διαφθορά σε διάφορες χώρες και υπάρχουν τέσσερις χώρες που πήγαν χειρότερα από ό,τι παλιότερα. Σχετικά με τα Ηνωμένα Έθνη, η εμπειρία μου με τα Ηνωμένα Έθνη είναι ότι δεν σου δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις ε, τους δικούς σου δημοσιονομικούς ελεγκτές αλλά νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να επιδιώξουμε με διάφορους τρόπους να υπάρξουν καλύτεροι έλεγχοι. Τώρα για τις εξωτερικές υπηρεσίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα γιατί υπάρχουν ορισμένες οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα. Ο Κωνσταντς ξεκινήσουμε στο τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων μετά το 2013, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα υπάρχοντα ταμεία. Βλέπουμε στο έγγραφο του ελεγκτικού συνεδρίου ότι εκεί που ζητούνται εξηγήσει είναι τα πολιετή γενικότερα προγράμματα και το πιο σοβαρό είναι το θέμα που αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη. Υπάρχουν ε, 13.000 ερευνητές οι οποίοι αρνούνται να συνεργαστούν στα προγράμματα της Ένωσης γιατί θεωρούν ότι είναι αντικείμενο ανεπαρκούς διαχείρισης. Και πολλοί πιστεύουν ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να επιστραφούν στα εθνικά κράτη για να γίνουν αντικείμενο καλύτερης διαχείρισης. και υπάρχουν και στην εκλογική μου περιφέρεια άνθρωποι που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα γι' αυτό γιατί έχουν προβλήματα εξ αυτού. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι αποτελεσματικότητα έχουν οι προσπάθειες που κάνουμε, γιατί στο τέλος κανένας δεν θα θέλει να πάρει τα χρήματα τα οποία εμείς θα προτείνουμε. Κωνσταντς, θέλω να αναφερθώ σε δύο σημεία, κύρια Πρόεδρε. Καταρχήν το θέμα της διαχείρισης των ταμείων. Ε, στην πολιτική συνοχή έχουμε δει στην πράξη ότι αντιμετωπίσαμε μεγάλες δυσκολίες για να εφαρμόσουμε τους κανόνες οι οποίοι είναι πολύπλοκοι και ποικίλουν κάθε φορά μεταξύ των ταμείων και των προγραμμάτων. Είχαμε τονίσει την ανάγκη να υπάρξει μια απλοποίηση, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε όχι μόνο και για, όχι μονάχα για απλούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής συνοχής, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε επίσης και ποιοι θα πρέπει να είναι οι κοινοί κανόνες οι οποίοι θα διέπουν το σύνολο των ταμείων, κοινωνικό ταμείο, περιβάλλον, προγράμματα έρευνας, εκπαίδευσης κτλ. Και φυσικά και το Ταμείο Συνοχής, ώστε να μπορούν να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι είναι κανόνες γενικής ισχύως, οι οποίοι είναι απλοί, είναι διάφανοι, είναι αποτελεσματικοί, ώστε να μην χρειάζεται κάποιος ο οποίος ζητά χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φορά να λειτουργεί με διαφορετικούς κανόνες. Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι της προβληματικής μας λοιπόν. Ξέρω ότι η Κομισιόν σκέφτεται για την απλοποίηση, αλλά είναι απαραίτητο και εμείς να τονίσουμε την ανάγκη να υπάρξει μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια και έχει δίκιο ο Γκέρον θα πρέπει να κάνουμε και ένα έλεγχο με γνώμονα το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών. Και έχουμε μια εμπειρία λοιπόν ήδη που έχει συσσωρευτεί. Πολλές φορές ένα πρόγραμμα έχει καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν ικανοποιεί αυτό το ελεκτικό συνέδριο, διότι δεν έχουν τηρηθεί ορισμένε διαδικασίες. Επίσης, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων και σχεδίων, φταίμε και εμείς ως ευρωπαϊκό όργανο όταν δεν προχωρούν αρκετά γρήγορα τα προγράμματα στην αρχή της περίοδου ζωής τους. Όταν ξεκινήσαμε νέα προγράμματα το 2007, υπήρχαν ήδη τον Ιούνιο του 2007 αρκετά λίγα προγράμματα τα οποία ήταν σε κατάσταση να λειτουργήσουν. Εκεί δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα οι περιφέρειες για να το βελτιώσουν. Και όταν τελικά όταν παίρνονται οι αποφάσει μόνο προ το τέλο του προηγούμενου έτου του 2006 για προγράμματα τα οποία πρέπει να εκτελούνται για το 2007, τότε και η ίδια η Κομισιόν δεν μπορεί να προετοιμάσει σωστά αυτά τα προγράμματα. Επομένω θα πρέπει και εμεί να παίξουμε το ρόλο μα μέσα στη διαδικασία στην απόφαση που μα δίδει η συνθήκη τη Λισαβόνα, ώστε να γίνονται, να λαμβάνονται εγκαίρω οι αποφάσει για τα προγράμματα αυτά. Αυτό θα βελτιώσει λοιπόν και την καμπύλη εφαρμογής για τα προγράμματα και σχέδια αυτά. Και επομένως δεν θα περιοριζόμαστε με το νησιν 2 ή νησιν 3, αλλά θα μπορεί να υπάρχει και μια επικάλυψη στο χρόνο των προγραμμάτων αυτών που θα βελτιώσει την εκτέλεσή τους. Ευχαριστώ, Derek Walt, Miguel Portus και θα κλείσει ο Σαλβαδόρ και δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητέ. Εγώ κλείσει τον κατάλογο για αυτό το θέμα. Okay, thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σχόλια. Πρώτον, για την ε, χαμηλό δίκτυ εφαρμογή, ιδιαίτερα για την πολιτική συνοχή και τα διαρθρωτικά. Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι υπεύθυνο για το μειωμένο δίκτυο εκτέλεση Φταίει η τα κράτη-μέλη, οι περιφέρειες, αυτοί που έχουν αναλάβει να εκτελέσουν τα προγράμματα, υπερβολικός έλεγχος των διαφόρων διαδικασιών. Βασικό αυτό το ερώτημα. Και σε ένα τμήμα του εγγράφου αναφέρεται στην κοινή διαχείριση και το έγγραφο λέει 11% περιθώριο λάθος. Ο ελεγκτής δηλαδή ουσιαστικά λέει ότι το 11% των κονδυλίων διατρέχουν κίνδυνο. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ λάθους και απάτης. Πρέπει να την κάνουμε αυτή τη διάκριση. Φυσικά τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε και μια νέα έκθεση και θα αναφέρεται μάλλον βελτίωση εκεί. Η ισορροπία που μας ενδιαφέρει είναι οι απλοποιημένες διαδικασίες γιατί όλοι συμφωνούμε ότι ένα τμήμα της λύσης είναι αυτό, αλλά χρειάζεται και υγιής δημοσιονομική διαχείριση. Στο παρελθόν έγινε προσπάθεια να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία. χάρη, η Κομισιόν εφαρμόσε ένα πρόγραμμα δράσης. Ας το δούμε. Ήταν επιτυχές. Την πέτυχε την απλοποίηση. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα όπου η Κομισιόν προσπάθησε να βελτιώσει την κατάσταση. Σε μερικέ περιφέρειες Φερρυπίν υπάρχουν συμβόλαια εμπιστοσύνη. Στην Ουαλία τα έχουμε αυτά τα συμβόλαια όπου το κοιτάει τα ε, συστήματα που ισχύουν οι Κομισιόν και αν είναι υγιή τότε δείχνει ευελιξία όσον αφορά την οικονομική διαχείριση. Δηλαδή επιτρέπει να εκτελούν ορισμένα πράγματα χωρίς να παρεμβαίνει περισσότερο πια η Κομισιόν. Ας δούμε λοιπόν μερικές από τις πρωτοβουλίες και τα παραδείγματα αυτά, να δούμε τι αποδίδει, τι αξίζει και να επεκτείνουμε τη χρήση αυτών περαιτέρω στο μέλλον. Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Μιγελ Πόρτους. Τρία ερωτήματα και μονάχα στα γρήγορα θα ήθελα να θέσω. Για τον κύριο Γκαρίγκα, εγώ πιστεύω ότι καταρχήν υπάρχει μια μεγάλη, μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ του ελέγχου σε προγράμματα γεωργίας και του ελέγχου σε προγράμματα της πολιτικής συνοχής. Πού βρίσκονται τώρα αυτές οι διαφορέ, Γιατί υπάρχουν τέτοιε διαφορές είναι το ερώτημα. <clears throat> Αυτό θα ήθελα να κατανοήσω. Το δεύτερο ερώτημα είναι πάλι για τον εισηγητή. Ο κύριος εισηγητή, αν μπορούσε να μας δώσει κάποια στοιχεία για το πόσο είναι, ποιο είναι το βάρος, ποιο είναι το τμήμα ενός, αν θέλετε, θελησιοκρατικού, βολονταριστικού προϋπολογισμού ε, που περιλαμβάνει και αυτά τα οποία ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, μήπως υπάρχει κάποια κίνηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οδηγεί σε υπερ εγγραφή κονδυλίων στον προϋπολογισμό που μετά φυσιολογικά δεν μπορούν να εκτελεστούν. Ένα τρίτο ερώτημα μέσα στις διαφορές που υπάρχουν για τους μηχανισμούς ελέγχου για τα διάφορα σχέδια και προγράμματα. θα μπορούσαν κάποιοι από αυτούς τους μηχανισμούς να κάνουν κάποια διάκριση μεταξύ προγραμμάτων που έχουν μικρές επενδύσεις και προγραμμάτων που έχουν μεγάλες επενδύσεις. Μήπως θα πρέπει να είναι διαφορετικές συνθήκες ελέγχου. <clears throat> Παραδείγματο χάρη, τα κονδύλια για την εξωτερική δράση, για την ε, ανάπτυξη. <clears throat> όταν γίνεται διανομή κονδυλίων σε μικρούς φορείς που είναι μη κυβερνητικοί, που παίζουν πάρα πολύ σημαντικοί φορείς για την ανάπτυξη, ένα μεγάλο μέρος του χρήματος <clears throat> πηγαίνει στην ανάγκη να κάνουν αυτοί οι οργανισμοί την απαραίτητη ε, λογιστική, να συντάξουν εκθέσεις, δηλαδή πηγαίνουν σε γραφειοκρατία τελικά όλα αυτά τα χρήματα. <clears throat> Ενώ σε προγράμματα που καταδαπανούν εκατομμύρια και εκατομμύρια ευρώ, φυσικά δεν είναι το ίδιο το, το άχθος της γραφειοκρατίας σε σχετικούς όρους όπως τα μικρά προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα να απαγορεύσω σε όλους τους συναδέλφους να ξαναπούν ότι θα είναι σύντομοι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να απογοητευόμαστε συνέχεια. Ο Σαλβαδόρ παρακαλώ για να κλείσει αυτή τη συζήτηση. Πάρα πολύ σύντομα. Γιατί θα ήθελα να μιλήσει και ο Επίτροπος. Ναι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις ε, συνεισφορές των συναδέλφων που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο για την εκπόνηση του εγγράφου αυτού που θα πρέπει να συντάξουμε. Να κάνω προς την αρχή κάποιες ε, παρατηρήσεις αυτοί που δεν θα τύχουν απάντηση τώρα θα δουν την απάντηση στην αναθεωρημένη μορφή του εγγράφου εργασίας. Στο παράτημα του εγγράφου αυτού, αν πάτε στη σελίδα 8, βλέπετε την εξέλιξη των πλεονασμάτων του προϋπολογισμού. <clears throat> Και υπήρξε ένα ερώτημα σε σχέση με την διάρκεια των δημοσιονομικών περιόδων, αν αυτό έχει κάποια σχέση με τον κύκλο λοιπόν. Το 2001, 2008 μάλλον υπήρχε μία, ένα υψηλό ποσοστό το 2007 υπήρχε μεγάλη επικάλυψη με το προηγούμενο ε, με τις προηγούμενες δημοσιονομικές προοπτικές, αλλά δεν επαναλήφθηκε αυτό το μεγάλο ε, πλεόνασμα. Και έτσι το 2007-2009 δεν βλέπουμε να υπάρχει μια αύξηση αυτού του πλεονάσματος. Βλέπουμε δηλαδή να υπάρχει και μια βελτίωση από την διαχείρι... για τη διαχείριση των πόρων τόσο από την Κομισιόν όσο και από τα κράτη-μέλη. Πάντα θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της απλοποίησης των διοικητικών ελέγχων και το έγγραφο σκέψης θα πρέπει να αντανακλά το επίπεδο εκτέλεσης σε επίπεδο πιστώσεων υποχρεώσεων και πληρωμών και επίσης να ξέρουμε τι είναι το καλύτερο για να εξασφαλίσουμε αυτήν την, ε, αυτήν την ε, εκτέλεση του μου. Το ερώτημα επίσης του αν πρέπει να κάνουμε έλεγχο σε σχέση με τη διαδικασία, με σχέση με το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η άποψη του Κοινοβουλίου μέχρι τώρα έχει σταθεί ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα και όχι στη διαδικασία. Και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την κοινή διαχείριση με μη κυβερνητικού οργανισμούς, με τον ΟΗΕ κτλ. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέσα στον έλεγχο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τις κοινέ της κοινή διαχείρισης ζητήσει έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων αυτών που πηγαίνουν σε διεθνείς οργανισμούς. Γιατί αυτό είναι τμήμα μια συμφωνία εμπιστευτικότητα που υπάρχει με του οργανισμού, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν τηρούμε ένα τμήμα τη της εντολής μας ως Επιτροπή που είναι ως ε, ελεγχτές του προϋπολογισμού που είναι ο έλεγχος όλων των πόρων του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης για την ιστορία, το ιστορικό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού έχουμε δει να υπάρχει έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εθνικών ελεγκτικών φορέων του και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και ξεκινάμε από μια βασική αδυναμία ότι τα ευρωπαϊκά <clears throat> όργανα έχουν ένα, νιώθουν ένα πανικό μπροστά στον κίνδυνο να υπάρξουν σφάλματα στη διαχείριση ακριβώς γιατί το Κοινοβούλιο στο παρελθόν είχε σταθεί πάρα πολύ στεναρό και αυστηρό σε σχέση με τα θέματα αυτά. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι θεωρούσαν ότι είχαν υπάρξει τεράστιες πολιτικές καταστροφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της έλλειψης επαρκούς ελέγχου και κάποια στιγμή πέσαν και κεφάλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγγνώμη. Αλλά φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να είναι η αρμόδια για τον έλεγχο, αλλά τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία διαχειρίζονται το 80% των πόρων. Ενώ η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Σούρε, εμείς προς το παρόν δεν έχουμε προτείνει μια μελλοντική λύση. Όσο δεν υπάρχει μια μελλοντική λύση, θα εξακολουθήσει αυτό το πρόβλημα. Επομένω, θα ήθελα να σα παρακαλέσω να σκεφτείτε λίγο περισσότερο για αυτό το σημαντικό θέμα, το οποίο θα μπορούσε να δώσει λαβή σε σημαντικέ προτάσει και για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ, λέει και η πρόεδρο. <clears throat> δεν θα μπορέσουμε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση τώρα αλλά θα έχουμε και πάλι ευκαιρίες να επανέλθουμε στο θέμα αυτό επί τη βάση του εγγράφου εργασίας. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημέρας διάταξης, το οποίο προβλέπει τη συζήτηση με τον κύριο Επίτροπο και χαίρομαι που ο κύριος Επίτροπος είναι μαζί μας και είναι έτοιμος να μας παρουσιάσει το review paper, το έγγραφο αναθεώρηση για τον προϋπολογισμό για να μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τι αλλαγές θα πρέπει να προέλθουν στην επόμενη περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών. Θέλω και πάλι να σας καλωσορίσω, κύριε Λεβαντόφσκι. Δεν ζητούμε την επίσημη παρουσίαση αυτού του εγγράφου, γιατί νομίζω ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι ήταν παρόντες όταν έγινε η παρουσίαση από την Επιτροπή του Εγγράφου Αναθεώρησης. Ίσως όμως θα μπορούσατε να κάνετε μια σύντομη παρουσίαση και στη συνέχεια θα δώσω την ε, δυνατότητα στις πολιτικές ομάδες με ένα εκπρόσωπό τους στη σειρά αριθμητική τους δύναμης να εκφράσουν τις απόψεις τους. Δεν χρειάζεται να είναι ο συντονιστής, αλλά όποιος είναι αρμόδιος για τα θέματα αυτά θα τους παρακαλέσω να λάβουν το λόγο, να σηκώσουν το χέρι τους και αν είναι ο, ο συντονιστής παρών θα ξέρω να τους δώσω το λόγο με τη σειρά. Αυτά για τη συνέχεια της ε, συζήτησης. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Thank you for your Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Δεν έχει περάσει πολύς χρόνος από την παρουσίαση αυτής της αναθεώρησης στην Ολομέλεια. Εσείς άμεσα εκλεγμένοι ήσασταν οι πρώτοι που ενημερωθήκατε γύρω από τα θέματα αυτά. Άκουσα μετά από δύσκολα σχόλια και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γκαρίγα. Είναι θέμα αριθμών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα παραρτήματα βέβαια. Στην ουσία κάνουμε μια εισαγωγή με κάποιες επιλογές δεν προκαταλαμβάνουμε πολιτικές αποφάσεις, αλλά κάνουμε κάποιες προτάσεις ε, για τους ίδιους πόρους, σαν παράδειγμα, που προκαλούν βέβαια αντιδράσεις. Υπάρχουν κάποιες νέες, ε, θα έλεγα, συζητήσεις από πλευράς του Συμβουλίου όλος περιέργως, ζητούν ότι κάποιοι ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το θέμα ε, των ιδίων πόρων. και από ό,τι φαίνεται υπάρχει τελικά μια κάποια δεκτικότητα για να συζητηθεί το θέμα των ιδίων πόρων στο Συμβούλιο. Το θέμα της διάρκειας, της χρονικής διάρκειας επίσης είναι ένα θέμα το οποίο ε, με απασχολεί. Η θέση του Κοινοβουλίου είναι πέντε χρόνια και είναι μια θέση η οποία μπορεί να τύχει υποστήριξης Το 5 συν 5 είναι κάτι το σχετικά υποθετικό γιατί προαπαιτεί ε, αναθεώρηση και προαπαιτεί επίσης και αποθεματικά και υποχρεωτικά αποθεματικά για τη δεύτερη περίοδο. Γιατί αν δεν υπάρχουν τα αποθεματικά προφανώς είναι θεωρητική συζήτηση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να αλλάξουμε τη σύνθεση ενός προϋπολογισμού και ενός κεφαλαίου. Και εδώ έχουμε επιλογές. Η μία είναι θα έλεγα ε, ρηξικέλευτη, σχεδόν επαναστατική, προσαρμοσμένη στους στόχους του 2020. Και η δεύτερη επιλογή είναι εδρεώνοντας κάποιους συγκεκριμένους τίτλους έτσι ώστε να έχουμε κάποια μεγαλύτερη ευελιξία. Επί της τώρα αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το θέμα της μόχλευσης σε τομείς όπως τα καινοτόμα μέσα. Στο σύνολο των επιτρόπων έχουμε μια ομάδα που ασχολείται με τα θέματα αυτά με στόχο να καταστήσουμε τη δυνατότητα αυτή λειτουργική. Σαν παράδειγμα τα πιθανά, αυτοί οι πιθανές συζητήσεις γύρω από τα ευρωομόλογα ή οι ευρωπαϊκές εγγυήσεις για ομόλογα. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν μέχρι τον επόμενο χρόνο. Υπάρχει πρόοδος λοιπόν σε σχέση με καινοτόμα μέσα, συνειδητοποιώντας βέβαια και τους περιορισμούς τους οποίους έχουμε. Κάποια άλλα θέματα που συνδέονται με τις συζητήσεις που κάνετε εσείς είναι ο δημοσιονομικός κανονισμός. Η Γκρέσλερ δεν είναι παρούσα να με ακούσει, έχει προσφέρει προς την κατεύθυνση αυτή. Η ετήσια προοπτική είναι ακριβώς μια κατεύθυνση συμβατή με αυτά τα οποία ακούστηκαν εδώ. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί ερευνητές δεν μπορούν πια την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία και θα ήθελα να υπάρξουν απλουστεύσεις ιδιαίτερα για μικρότερα ποσά. Όλες αυτές οι προσπάθειες ε, ε, βαδίζουν θα έλεγα παράλληλα και οδηγούν στην επεξεργασία του κεντρικού προβλήματος. Διάρκεια του προϋπολογισμού, σύνθεση του προϋπολογισμού, απλούστευση του δημοσιονομικού κανονισμού, καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, εκ νέου συζήτηση για τους ιδίους πόρους, Όλα αυτά αντικατοπτρίζουν την κατάσταση όπως υπάρχει σήμερα και όπως αναγνωρίζεται και από εσά εδώ στο Κοινοβούλιο και από τα κράτη-μέλη σχετικά με τη μορφή θα έλεγα και το περιεχόμενο της πολιτικής συνοχής. Υπάρχουν τάσεις που κρίνουν ότι η συνοχή αυτή θα πρέπει να είναι εδαφική τοπική και όχι γενικότερα να αντιμετωπίζεται ευρωπαϊκά. και πρέπει να δούμε και ποιο είναι όχι η ουσία μόνο, αλλά η θέση της αγροτικής πολιτικής. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι η τάση για μειούμενες διαστάσεις της κοινή αγροτικής πολιτικής είναι κάτι το οποίο θα προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις από αρκετές κυβερνήσεις και κοινοβούλια που αντιδρούν γενικά στην προσωπική κατά τα άλλα διατύπωση των προτάσεων. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο, είμαι περισσότερο εδώ για να δώσω απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ακούω τα σχόλιά σας, γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση ιδιαίτερα αποφασιστική θα έλεγα, στον τομέα ιδιαίτερα της πολιτικής συνοχής και της αγροτικής πολιτικής. Περιμένουμε να έλθουν πολύ σημαντικά έγγραφα. Ήδη τον Νοέμβριο θα έχουμε στη διάθεσή μας κάποια πρώτα στοιχεία. Νομίζω ότι όλα αυτά θα επηρεάσουν τις ανακοινώσεις της Επιτροπής και για την ε, Γεωργία και για την πολιτική συνοχή στον Ιούνιο του 2011. Έχουν ήδη εγγραφεί 7 για τις πολιτικές ομάδες. Εν πάση περιπτώσει θα πάρουν το λόγο 7 συνάδελφοι και μετά στους υπολείπους συναδέλφους θα δώσω το λόγο όταν το ζητήσουν. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για μια ακόμη φορά να είστε σύντομοι. Ο κύριος Μπέγκε θα μιλήσει πρώτος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την ε, θετική του εισαγωγή, όπως είχα ήδη την ευκαιρία να το πω και στην Ολομέλεια. Το έγγραφο αυτό δεν περιλαμβάνει όλα όσα θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχε εκφράσει ήδη από το 2006 και στα πλαίσια των συνδιαλλαγών και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων συζητήθηκαν πολλά θέματα και αυτό φαίνεται στο ενδιαφέρον περιεχόμενο αυτής της πρότασης η οποία όμως επαναλαμβάνω δεν ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτά τα οποία είχαμε στο νου μας σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απλούστευση, βελτίωση, καινοτομίες, όλα αυτά είναι απαραίτητα αν θέλουμε να απαλλαγούμε από την κόκκινη κάρτα την οποία μας είχε σηκώσει το ελεγκτικό συνέδριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί μας με θάρρος έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε σε κάποιες μεταρρυθμίσεις χωρίς αυτό να κλονίσει βέβαια την αρχιτεκτονική του δημοσιονομικού ελέγχου γενικότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι σε ορισμένους τομείς παρά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν υπάρχει μια δυνατότητα να βρεθούν κάποια επιπλέον ποσά. Για τους ιδίους πόρους τώρα. Το θέμα είναι πώς υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν σωστότερα ανακατηγορία. Να ξεκινήσω λοιπόν να μείνω λίγο στους ιδίους πόρους. Την Τρίτη ήμουνα στο Βερολίνο και συζητούσαμε συναδέλφους από την Ομοσπονδιακή Βουλή και είπα συνάδελφοι κοιτάξτε τι λέει η συνθήκη. Λέγει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από ιδίου πόρους για να χρηματοδοτήσει διαφορετικά ε, σημεία του προϋπολογισμού. Όποιος θέλει να σέβεται τη συνθήκη και το κοινοβούλιο μας πρώτο θα πρέπει να ασχοληθεί ε, με το θέμα των ιδίων πόρων. Εγώ δεν θα ήθελα να προκαταλάβω τα αποτελέσματα της συζήτησης αλλά θα ήθελα απλά να ζητήσω να σεβαστούμε τη συνθήκη. Υπάρχει λοιπόν συζήτηση και από τη συζήτηση αυτή θα βγουν ορισμένα τελικά συμπεράσματα. Όλες αυτές οι δυνατότητες λοιπόν θα πρέπει να ζυγιστούν και να ληφθούν υπόψη και ίσως θα χρειαστεί να αλλάξουμε κάποιες κατηγορίες εσόδων προς όφελος άλλων Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συνένεση στο τέλος για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Δεύτερον θα ήθελα να πω η Κομισιόν μιλάει στο έγγραφο αναθεώρησης για μια μεγάλη πλειάδα προοπτικών σε επίπεδο πολιτικών αυτών. Σωστό. Αλλά αυτό δεν πρέπει να αφορά μονάχα την πολιτική της Ευρώπης 2020 και αυτά που θέλουμε να πετύχουμε τώρα, αλλά και τη σχέση της πολιτικής προϋπολογισμού με την νομοθετική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα είπε ο κ. Επίτροπος, θα μειώσουμε τα αγροτικά ποσά και θα αυξήσουμε τα, τα θέματα της ε, πολιτικής συνοχής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως έχει πει ότι πρέπει να διατηρηθεί το επίπεδο των αγροτικών δαπάνων. Δεν μπορείτε εσείς σε ένα έγγραφο ή μη να πείτε ότι θα μειωθούν οι άμεσες πληρωμές χωρίς να λέτε από την άλλη μεριά ποια θα είναι η συνέπεια για το, για εισόδημα των ε, γεωργών και συγχρόνως να προχωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διμερείς συμφωνίες με χώρες όπως ο Καναδάς που έχουν μια προστατευτική λειτουργία μέσα στα πλαίσια της αγροτικής πολιτικής. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δεχτούμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει ίσως να σκεφτείτε καλύτερα και να συνοηθείτε καλύτερα με τις άλλες γενικές διευθύνσεις για να έχετε μια συνεκτική πρόταση. Γιατί αυτό το οποίο έχουμε ενώπιον μας αυτή τη στιγμή δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το θέμα τώρα της συνέχειας, νομίζω ότι εδώ το θέμα της χρηματοδότηση των υποδομών είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί στην περίπτωση αυτή είτε έχουμε δανειοδοτήσεις δανειοληψίες και οποιασδήποτε άλλες ε, δραστηριότητες, θα πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια συνέχεια στα σχέδια που έχουν να κάνουν με δημιουργία ε, υποδομών. Δεν πρέπει φυσικά αυτό να όρισε να σημάνει να σημαίνει ότι όλη αυτή η διαδικασία ξεφύγει από τα χέρια των ευρωπαϊκών θεσμών και θα γίνεται εκτός του έλεγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε όλες αυτές τις δραστηριότητες και νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό να γίνει παραγωγός χάρη στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και σε προγράμματα όπως το Γαλιλαίος και το ΙΤΕΡ θα ήταν απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει στην διαδικασία τροποποίησης διαχείρισης αυτών των ε, φορέων και επίσης να ξέρουμε ποια είναι η άποψή μας σε σχέση του Κοινοβουλίου, δηλαδή για τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα του ευρωπαϊκού, ε, του ευρωπαϊκού χώρου και εάν ναι, όχι κάθε φορά να μας αλλάζετε τις προτεραιότητες όταν έχετε η διαδικασία του προϋπολογισμού και να λέτε ναι χρειαζόμαστε και άλλα ποσά εδώ γιατί προήλθε ένα πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας σαφής τρόπος αντιμετώπισης. Μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχει ανάγκη ιδιαίτερων κανονισμών αλλά θα πρέπει όλη αυτή η διαδικασία να γίνεται με έναν τρόπο που θα είναι σαφέστερο σε επίπεδο ε, προϋπολογισμού. Νομίζω θα ήταν πολύ θετικό εφόσον μιλάμε για τα θέματα αυτά να σκεφτούμε τι σημαίνουν αυτά τα διαφορετικά υποδείγματα τα οποία ακολουθούμε. Η παράταση κατά τέσσερα χρόνια ξέρουμε ότι μια διάρκεια ζωής πέντε ετών για τα σχέδια και τα προγράμματά μας μπορεί να έχει νόημα μόνο αν παραμείνουν τα πράγματα όσοι έχουν σήμερα. Δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Αν μιλάμε για το 5 συν 5 σε διάρκεια, ίσως θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα πιο ισορροπημένο πακέτο ε, που θα προέρθει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που δεν θα έχει σαν αποτέλεσμα κάθε πέντε χρόνια να πρέπει να παίζουμε μπουνιές για το ποιες θα είναι οι δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτό μου σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και πιο στερεές δομές για το μέλλον. Θα πρέπει όχι απλώς να κάνουμε μια επιδερμική μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού, αλλά θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει πλήρως στην ε, λειτουργία του προϋπολογισμού και να υπάρχει η δυνατότητα ευκαμψίας του προϋπολογισμού για να υπάρχει αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, νέων αναγκών που μπορεί πριν απο 2 2-3 χρόνια να μην είχαν προβλεφθεί. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει αποδεκτό ένα τέτοιο μοντέλο. Πρέπει να μιλήσουμε, να συζητήσουμε για μοντέλα, αλλά σε όλα τα μοντέλα μαζί με την ευκαμψία είναι απαραίτητη και η δημοκρατική μονομιμοποίηση και ο έλεγχος. Μόνο με αυτή τη βάση μπορούμε και δίνω απόλυτο δίκιο <clears throat> στον Έλλες. Μόνο έτσι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες και ποιες είναι οι υποκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να δώσουμε την έγκρισή μας. Και πρέπει αυτό να το κάνουμε μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι την έγκριση του προπολογισμού για να μπορέσουμε να δούμε και ποιο ακριβώς μοντέλο θέλουμε να επιλέξουμε. Ευχαριστώ <clears throat> η κυρία Γκάρδια Σαμπάλ για, τις, για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λεβαντόσκη. Το πρώτο το οποίο ήθελα να σας πω είναι ότι το έγγραφό σας αυτό με, μου δημιουργεί μια μικρή σύγχυση. Γιατί αυτό δεν είναι μια τροποποίηση του τωρινού δημοσιονομικού πλαισίου, όπως ζήτησε η Επιτροπή Προϋπολογισμών και όπως είχατε δεσμευτεί να πράξετε. Λέτε ότι ούτε είναι και μια πρόταση για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, οι οποίες θα πρέπει ούτως ή άλλως να εξεταστούν στη συνέχεια, λέτε ότι είναι απλώς ένα έγγραφο που περιέχει διάφορες εναλλακτικέ λύσεις. Δεν ξέρω τι να το κάνω αυτό το έγγραφο. Δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένετε από εμά να κάνουμε με αυτό το έγγραφο. Δεν είναι μια πρόταση. Όλα αυτά είναι γραμμένα σε υποθετικό χρόνο και σε υποθετικό ύφος. Δεν είμαι σίγουρη λοιπόν ότι αυτό είναι τμήμα της συζήτησης που κάνουμε σήμερα στην Επιτροπή Σούρε Μιλάτε για συνοχή, μιλάτε για κοινή αγροτική πολιτική, μιλάτε για ένα νέο κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Όλα αυτά είναι συζητήσει που θα πρέπει να κάνουμε στην Επιτροπή μας και εξάλλου γι' αυτό υπάρχει η Επιτροπή Σούρε για να δούμε πώς θα έπρεπε να είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι μορφή πρέπει να αναλάβουν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα μπορέσουμε να τα καλύψουμε όλα αυτά και να τα ενσωματώσουμε στις επερχόμενες δημοσιονομικές πολιτικές, προοπτικές. Ξεκινάτε λοιπόν Φύγετε θέματα τα οποία έχουν μεγάλη εμβέλεια και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά δεν μπορούμε εμείς τώρα να συζητήσουμε αυτό το οποίο λέει το έγγραφό σας, γιατί τότε αυτό θα σήμαινε ότι είχαμε κλείσει το έργο της Επιτροπής μας. Δηλαδή θα περιοριζόμασταν να εκφράσουμε άποψη για το έγγραφό σας και θα έχει τελειώσει η εργασία μας. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ λοιπόν παρά το γεγονός ότι δεν ξέρω ακριβώς από πού να πιάσω αυτό το έγγραφο, θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια για ορισμένε πτυχέ του εγγράφου αυτού. Όπως σας ε, είπα στην αρχή, εμείς θέλαμε ένα έγγραφο για την μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών προοπτικών, επειδή έχει τεθεί σε εφαρμογή η Συνδίκη Λισαβόνα, επειδή έχουμε ενώπιον μα τη στρατηγική τη Ευρώπη για το 2020 και ξέρουμε όλοι ότι δεν έχουμε αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε αυτή την πολιτική. Κάτι το οποίο εσεί δεν θίγετε καθόλου στο έγγραφό σα. Επομένω, αυτό δεν αντιστοιχεί σε αυτά που ζητήσαμε. Και είναι ακριβώ το θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή Σούρε. Κάτι ακόμα το οποίο μου φαίνεται πολύ παράξενο. Μιλάτε για την ευκαμψία, την ευελιξία, τη σημασία που έχει η ευκαμψία. Και εμείς ως Επιτροπή Προϋπολογισμού το έχουμε τονίσει αυτό. Αλλά η σημασία της ευελιξίας είναι να είναι κάτι το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς, να υπάρχουν κάποια εργαλεία, να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ε, τροποποιήσεις στις δημοσιονομικές πολιτικές. Το πρόβλημα είναι ότι η ευελιξία υπάρχει θεωρητικά, αλλά δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Και κάτι ακόμα που μου φαίνεται πολύ σημαντικό και αυτό είναι κάτι το οποίο τονίζει ιδιαίτερα η σοσιαλιστική ομάδα. Το θέμα των ιδίων πόρων. Σε κάποιο σημείο θίγεται βέβαια στο εγγραφό σας το θέμα των ιδίων πόρων και το Συμβούλιο φαίνεται, τουλάχιστον φαίνεται, έτοιμο να συζητήσει για τα θέματα αυτά. Όχι να φτάσει σε μια συμφωνία, αλλά να το συζητήσει. Και στο εγγραφό σας αναφέρεται κάποιες ιδέες δυνητικές για ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. όλα αυτά δεν είναι ακόμα απτά και συγκεκριμένα. Μου φαίνεται όμως παράξενο ένα θέμα που έχει συζητηθεί τόσο πολύ όπως είναι ο φόρος στις ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές και το οποίο το είχε υποστηρίξει η σοσιαλιστική ομάδα και είχε παρουσιάσει και τροπολογίες στον προηγούμενο προϋπολογισμό μου κάνει εντύπωση που δεν εμφανίζεται καθόλου αυτό το έγγραφο, που δεν υπάρχει καμία αμνία και μιλάτε για συνέργεια μεταξύ του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και των εθνικών προϋπολογισμών, της κρίσης, της λιτότητας, της ανάγκης να βελτιωθούν οι δαπάνες και η ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία. Και αυτό με το θέμα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Μόνο επειδή έχουμε μία κρίση, <clears throat> μόνο επειδή περνάμε δύσκολες στιγμές θα πρέπει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των δαπανών μας και να δώσουμε ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία. Όχι, αυτό θα πρέπει να ισχύει και σε περίοδους κρίσης και σε περίοδους παχαίων αγελάδων. Γιατί το να έχουμε καλύτερη διαχείριση μόνο στην περίπτωση μιας κρίσης, αυτό μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι σε άλλες περιπτώσεις δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, δεν πρόκειται να σχολιάσω γιατί θέλω να ακούσω και τι λένε οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Αλλά σας ξαναλέω κύριε Λεβαντόσκη, τι ακριβώς θέλετε να κάνουμε με το έγγραφό σας, πώς θέλετε να το αντιμετωπίσουμε σαν Επιτροπή. Γιατί από τη μία πλευρά θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν κομμάτι της λειτουργίας της Επιτροπής μας και να σας ευχαριστήσουμε για τις ιδέες σας. Από την άλλη μεριά μπορεί να το αντιμετωπίσει κανείς ότι είναι μια προσπάθεια παρέμβαση στο έργο της Επιτροπής μας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Αλλά από τη δική σας πλευρά ως Κομισιόν τι επιζητείτε με το έγγραφο αυτό. Ähm, Ευχαριστώ, Έντεν. Έντνα. Ίσως θα μπορούσε η Επιτροπή να ονομάσει αυτό το έγγραφο αναθεώρησης έγγραφο σκέψης. Και τότε δεν νομίζω ότι θα υπήρχε πρόβλημα με να το συμπεριλάβουμε στην, ε, στον προβληματισμό μας. Ο Κάλλη έχει το λόγο. Καταρχάς ξεκινώντας θα ήθελα να ξεκινήσω, να αρχίσω με τα θετικά. Πράγματι θέλουμε όλοι να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση για τους ιδίους πόρους. Και μας ικανοποιεί το γεγονός ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει προς την κατεύθυνση αυτή. Και οι συνάδελφοί μου από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα θα ήθελαν να πούμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις uh, place. So, so this is a very good part of the document. Και σε όλες τους, τις ιδέες για φόρους που θα μπορούσαν να είναι γενικά θεμητές νομίζω. Το ίδιο επίσης και για τα ευρωομόλογα. Πολλές ιδέες μπορούν εδώ να γίνουν πραγματικότητα για τη χρηματοδότηση της Ευρώπης. Υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία λοιπόν προς συζήτηση και επίσημα πλέον. Θα πρέπει επίσης να συμφωνήσω με τον προηγούμενο συνάδελφο ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κατανοήσει κανείς τον ρόλο που έχει αυτό το έγγραφο. Ένα από τα έγγραφα τα οποία μας μοιράστηκε λέγεται «Ε, μαθήματα που μπορεί να πάρει κανείς από τον αυριανό προϋπολογισμό και αναρωτιέμαι τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο δικό μου κόσμο το αύριο είναι το 2011, το 2013, 2014 και πάει λέγοντας. Έχουμε συμφωνήσει σε μια πολύ φιλόδοξη πολιτική και έχουμε θα έλεγα γενικότερα πολύ φιλόδοξους στόχους για τα επόμενα χρόνια και αυτό κανονικά θα έπρεπε να αντικατοπτρίζεται στο έγγραφο το οποίο μας έχει δοθεί. Πώς θα μπορέσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας διαβεβαιώσει ότι η στρατηγική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί τα επόμενα δύο χρόνια, τρία χρόνια πριν περάσουμε στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, να προχωρήσουμε. Πριν φτάσουμε στο 14 έχουμε το 13, έχουμε το 12, έχουμε το 11. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το 30%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάρα πολύ σωστά λέγει ότι οι κάποιες μετακινήσεις στο εσωτερικό του προϋπολογισμού μπορούν να γίνουν ένα αλλά σε περιορισμένο πλαίσιο και με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. όταν υπάρχουν αλλαγές στις συνθήκες και τα λοιπά. Προφανώς και απαιτείται να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν το 2011, 12 και 13, όχι μόνο μετά το 2014. Πολλές ιδέες ε, προτείνονται για τις παρούσες δημοσιονομικές προοπτικές και οι περισσότεροι από εμά θα συμφωνήσουμε με το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού, αλλά το πιο προβληματικό είναι ότι δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φανταστούμε ποιες είναι οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ορισμένα θέματα. Δεν διαφωνεί κανείς με αυτά τα οποία προτείνονται, αλλά θέλουμε πολύ πιο συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα δουλέψουμε τα επόμενα τρία χρόνια. Εγώ δεν νομίζω ότι θα επιβιώσουμε βλέποντας ε, ποιο τμήμα ε, του προϋπολογισμού του σημερινού στηρίζει τη στρατηγική του 2020. Έχουμε ένα ποσοστό το οποίο φαίνεται ικανοποιητικό, αλλά το ποσοστό αυτό δεν δείχνει τις αλλαγές στα δημοσιονομικά μας. Αφορά τον παρόντα προϋπολογισμό. Δεν αναφέρεται στο τμήμα του προϋπολογισμού που μπορεί πράγματι να εφαρμοστεί για την εξυπηρέτηση της στρατηγικής 2020 και τι αλλαγές θα πρέπει επίσης να κάνουμε στον προϋπολογισμό για να υπηρετήσουμε τη στρατηγική αυτή καλύτερα. Δεν βρίσκω μέχρι τώρα απαντήσεις ούτε σε αυτό το έγγραφο ούτε στα υπόλοιπα έγγραφα τα οποία έχει δώσει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό λοιπόν το έγγραφο αυτό, θέλουμε όμως περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Καρλ. Στον κατάλογο έχω τους πράσινους. Ο Ράινερ Μπιουτικόφερ ήθελε να λάβει το λόγο. Μιλάει ως Μπουτικόφερ ή ως Πράσινος. Αν μιλήσει για τους Πράσινους, μπορώ να τους δώσω το λόγο. Αλλιώς πρέπει να το δώσω το λόγο στην Χέλγα. Ως Πράσινος θα μιλήσω. Αλλά πρώτα οι κυρίες. Προηγούνται οι κυρίες, λέει ο κύριος Μπουτικόφερ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να υπάρξει διαμάχη. Εντάξει, θα μιλήσω εγώ για τους πράσινους λέει Χέλγα. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για το έγγραφό σας. Το οποίο είναι πράγματι περισσότερο σαν ένα έγγραφο σκέψης και όχι ένα έγγραφο αναθεώρησης για το 2012-2013. Εδώ θέλω να σας επικρίνω και γι' αυτό θέλω να θέσω και ένα πολιτικό ερώτημα. Βλέπω να υπάρχουν πολλές καλές προτάσεις στο έγγραφο αυτό, αλλά υπάρχουν και δυσκολίες με τις λεπτομέρειες. Εγώ προηγουμένως όμως θέλω να σταθώ στο στρατηγικό ερώτημα. Βρισκόμαστε τώρα σε διαδικασία διαβούλευσης με το Συμβούλιο. Και το Κοινοβούλιο έθεσε τα λεγόμενα 7 μεγάλα θέματα στο ψήφισμά του. Και θεωρείται μέσα στο πλαίσιο αυτό ότι ο προϋπολογισμός του 2011 θα είναι μεταβατικός προϋπολογισμός, αλλά από το 2012 θέλουμε να υπάρχουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις και όχι το Συμβούλιο να διατηρήσει την τωρινή κατάσταση μέχρι το 2014 χωρίς να υπάρξει καμία ποιοτική τροποποίηση στον προϋπολογισμό. Ποιος είναι ο δικός σας πολιτικός ρόλος κύριε Επίτροπε, και πού βρισκόσαστε μεταξύ των συμφερόντων του Συμβουλίου και των δικών μας. Πού θέλετε να κινηθείτε μέσα στο, στα πλαίσια του εγγράφου σας και ποια είναι η άποψή σας. Θέλετε να υπάρξουν κάποιες αλλαγές το 2014 μονάχα ή θέλετε να γίνουν και προηγουμένως. Αυτό είναι ένα σαφές πολιτικό ερώτημα. Ποιος είναι ο πολιτικός λοιπόν πυρήνας αυτού του εγγράφου θα θέλαμε και από πότε θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτές οι τροποποίησεις. Γιατί όλα αυτά θα έχουν μεγάλη σημασία για το δεύτερο τμήμα της ε, περίοδου δημοσιονομικών προοπτικών. Εκτός αν θέλετε να γίνουν αυτές οι αλλαγές μονάχα μετά το 2014. Μετά είναι και το ερώτημα που έθεσε η συνάδελφος από τους ε, σοσιαλδημοκράτες. Τι θα γίνει με τη στρατηγική του 2020, μήπως χρειάζονται και ποιοτικά νέες ιδέες για το πώς θα μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε την πολιτική μας οικονομικής ανάπτυξης και την κάνουμε πιο ε, αηφόρο επίσης, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο περιβάλλον, στην εκπαίδευση κτλ. Μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε πριν από το 2014. Ποιος είναι ο πολιτικός ρόλος της Κομισιόν σε αυτό το, ε, το εγχείρημα. Θέλετε εσείς λοιπόν να ξεκινήσουμε πιο νωρίς ε, στο συμφέρον της Ευρώπης ή πρέπει να χάσουμε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι το 2014. Αυτό είναι το ερώτημά μου λοιπόν προς εμάς και θα ήθελα πολύ να το απαντήσετε. Ευχαριστώ τους πράσινους. Η ομάδα των συντηρητικών παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το ότι έχουμε το έγγραφο από την Κομισιόν, αυτό είναι θετικό, είναι ένα σημαντικό έγγραφο. Βρισκόμαστε βέβαια σε μια φάση συζήτησης και είναι χρήσιμη συνεισφορά στη συζήτηση αυτό. Θα ήταν όμως πατάλιο χρόνο να συζητάμε μόνο τους ιδίους πόρους. Βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Σαν να μην υπάρχει διάθεση να γίνει συζήτηση για μια νέα α, διανομή, κατά κάποιο τρόπο αναδιανομή των εσωτερικών πόρων πώς θα δαπανώνται τα χρήματα αυτά μεταξύ των κρατών μελών και των Βρυξελών. Δεν ξέρω λοιπόν αν αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε αυτό τώρα. Εκεί που έχω μερικές αμφιβολίες είναι από τη μια μεριά η προστιθέμενη αξία και από την άλλη μεριά οι πιο φτωχές περιφέρειες. Η υποστήριξη των πιο φτωχών περιφερειών διατυπώνεται με μια γλώσσα που δεν είναι πολύ εγωιστική. Δηλαδή η υποστήριξη των πιο φτωχών περιφερειών είναι η πιο καλή έκφραση του τι σημαίνει τη προστιθέμενη αξία στην Ένωση. Διότι έτσι θα μπορούν να ωφεληθούν πλήρω από την ενιαία αγορά και για να ωφεληθούν, αν ωφεληθούν μάλλον, αυτό θα ήταν ένα τεράστιος παράγοντας που θα μας βοηθούσε όλους μας να βγούμε από την κρίση. Η κοινή αγορά είναι χρήσιμη για όλους μας και οι χώρες που πληρώνουν και οι χώρες που λαμβάνουν τους πόρους, τα ωφέλη, τα βλέπουμε αυτά με βάση όλους τους δείκτες και παραμέτρους που έχουμε στα χέρια μας για τα τελευταία χρόνια στην μακροκλίμακα και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την πολιτική συνοχή, Αυτό το καταθέτω ως επικριτικό σχόλιο σχετικά με το περιεχόμενο του εγγράφου. Το έγγραφο αυτό καθεαυτό είναι ευπρόσδεκτο. Ähm, Ευχαριστώ η Γκουε, ο Μίγκελ. Δεν θα κάνω τώρα εκτενείς παρατηρήσεις για το ότι αυτό είναι έγγραφο σκέψη περισσότερο από έγγραφο αναθεώρησης θα το εξετάσω σε επίπεδο ουσίας σαν στοιχείο σκέψης. Έχω μια πρώτη αμφιβολία εδώ, η οποία είναι η Υπάρχει μια εγγενής, μια υποβόσκουσα κατά κάποιο τρόπο επιλογή σε αυτό το έγγραφο που λέει ότι σε επίπεδο προϋπολογισμού το βασικό είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα. και τα λεγόμενα νέα μέσα, τα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης θα πρέπει να αφιερωθούν στη χρηματοδότηση ειδικών σχεδίων, συγκεκριμένων σχεδίων. Δηλαδή, μιλάμε για ένα προϋπολογισμό της ίδιας τάξης μεγέθους και χωριστά άλλους διευρυμένους πόρους για συγκεκριμένα μονάχα σχέδια. Και εδώ έχω την πρώτη αμφιβολία για αυτό το υπόδειγμα το οποίο παρουσιάζεται. Είναι ένα σωστό μοντέλο αυτό. Έχω πολλές αμφιβολίες για κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε σημαντική ε, αύξηση σε αποδοτικότητα και πρέπει να το επιζητήσουμε αυτό, αλλά αμφιβάλλω για το αν μια μεγαλύτερη παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέδια τα οποία θα οδηγήσουν σε οικονομική μεγέθυνση και θέσεις εργασίας μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει μονάχα μέσα από τα νέα μέσα χρηματοδότησης. Υποστηρίζω αυτά τα σχέδια, τα ευρωομόλογα παραδείγματος χάρη, αλλά όπως είπε και ο κύριος Μπέγκε προηγουμένως, τα καινοτόμα αυτά μέσα θέτουν ένα πραγματικό πρόβλημα δημοκρατικού ελέγχου. Πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να έχουμε εμεί κάποιο έλεγχο στους μεγάλους φορείς <clears throat> οι οποίοι θα αναλάβουν τη σκητάλη, θα αναλάβουν την πραγματική διαχείριση της χρηματοδότησης αυτών των μεγάλων σχεδίων που αναφέρει η Κομισιόν. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω. Και ακολουθεί τώρα μία παρατήρηση σε σχέση με τα δεκαετή δημοσιονομικά πλαίσια με ενδιάμεση αναθεώρηση στα πέντε χρόνια με την προηγούμενη εμπειρία που έχουμε συσσωρεύσει, πώς μπορεί να μας εγγυηθεί η Κομισιόν <clears throat> ότι τα κράτη-μέλη θα δεχτούν να κάνουν ενδιάμεσες αναθεωρήσεις στη μέση της δεκαετούς περίοδου. Γιατί ξέρουμε ήδη από το τωρινό χρηματοοικονομικό, δημοσιονομικό μάλλον πλαίσιο, όπου τα κράτη-μέλη έχουν συνάψει μια συμφωνία, μια διαθεσμική συμφωνία με το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν <clears throat> να γίνει μια ενδιάμεση, ενδιάμεση αναθεώρηση. Και όταν φτάνει η στιγμή αυτή για την αναθεώρηση λένε δεν θέλουμε και θα, θα κάνουμε τίποτα. Αν προτείνω να περάσουμε λοιπόν <clears throat> σε επίπεδο σχεδιασμού 10 ετών όλα τα προβλήματα της ενδιάμεσης αναθεώρησης θα πρέπει να έχουν να συνοδεύονται από τεράστιες εγγύησεις γιατί αλλιώς θα έχουμε δημοσιονομικές προοπτικές που θα είναι ένας στενός κορσές 10 ετών που δεν θα έχει δυνατότητα να ανταποκριθεί στις πραγματικότητες της σύγχρονης που είναι η τεράστια αβεβαιότητα σε οικονομικό επίπεδο. Πώς θα καταφέρει λοιπόν ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αβεβαιότητες στον οικονομικό στίβο. Εγώ δεν νομίζω ότι το έγγραφό σας απαντά σε αυτό το ερώτημα. Τρίτο ερώτημα. Το κείμενο αυτό περιέχει πολλές σιωπές. Εγώ άκουσα τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόζο, να μιλάει πολλές φορές επανειλεμμένα να υπάρξει, για την ανάγκη να υπάρξει μια συμπληρωματική κοινωνική πολιτική, συμπληρωματική των πολιτικών που ακολουθούνται από τα κράτη-μέλη. Εγώ δεν, μπορώ, να συμφωνήσω περισσότερο με αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μπαρός. Αλλά αυτό δεν το βλέπω να αντανακλάται σε αυτό το κείμενο και αναρωτιέμαι γιατί δεν περιέχετε στο κείμενό σας όταν έχετε τόσα άλλα πράγματα που αναφέρετε. Και ένα δεύτερο ερώτημα λίγο πιο πολύπλοκο που θέλω να θέσω. Η Ευρώπη έχει μπει ήδη σε μία πορεία απόκλησης των χωρών που την απαρτίζουν. Ήδη μέσα στη ζώνη του ευρώ υπάρχει μια διαρθρωτική απόκληση στις οικονομικές πολιτικές των χωρών στην ζώνη του ευρώ. Και ξέρουμε ότι οι πολιτικές συνοχής δεν καταφέρνουν να αλλάξουν αυτή την πορεία απόκλησης μέσα στην οποία έχει μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κρίση οικονομική οξύνει όλα αυτά τα θέματα. Επομένως το ερώτημα το οποίο θέτω είναι το εξής με ποιο τρόπο μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο απόκλησης πολιτικών και το σενάριο αυτό της απόκλησης των πολιτικών είναι πολύ πιθανό θα συνεχίσει, πώς σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει την κοινωνική διάσταση μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Γιατί στο παρελθόν λέγαμε ότι αν με την πολιτική συνοχή επιληθούν τα προβλήματα θα υπάρχουν θετικές ε, επιπτώσεις στο κοινωνικό επίπεδο, αύξηση των προσώτων, μεγαλύτερη απασχόληση κτλ. Τώρα όμως όχι. Τώρα φαίνεται ότι οι πολιτικές συνοχής δεν είναι επαρκείς για να αντιμετωπίσουν την επιδείνωση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πολύ πολύ να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές ανισότητες μέσα σε κάθε συγκεκριμένη χώρα, αλλά όχι τις κοινωνικές ανισότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής, η κυρία Ανδρία, αν έχει το λόγο, <clears throat> για τη δική της πολιτική ομάδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει μια κάποια σύγχυση σχετικά με το στόχο αλλά και το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι αυτό δείχνει ότι δεν καταλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι χρειάζεται για να υπάρξει ένας ουσιαστικός και αποτελεσματικός προϋπολογισμός. Αυτή η ανησυχία μου είναι η ίδια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν λοιπόν δύο προβλήματα. Ένα από αυτά το έχουμε αντιμετωπίσει επανειλημμένα. Τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξουν για τον προϋπολογισμό του 2011 ένα επιπλέον ποσό 300 εκατομμύρια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει μια διορθωτική επιστολή για μείωση του προϋπολογισμού αυτού, του τμήματος αυτού για το 2010. Ε, αυτό είναι αυτό που θα ονόμαζα αναποτελεσματικός προϋπολογισμός. Ποιο είναι το παιχνίδι της Κομισιόν. Αναρωτιέμαι καταλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σύνδεσμο ανάμεσα σε ένα ανεπαρκή προϋπολογισμό και την έλλειψη κανονικότητας στην οποία ανοιχνεύει το ελεγκτικό συνέδριο συστηματικά από τον ένα χρόνο στον άλλο. Αν αυτές οι ελλείψεις κανονικότητας οδηγούν σε απάτες είναι θέμα προσυζήτηση, αλλά στα Ταμεία Συνοχής, σαν παράδειγμα στο Ταμείο Συνοχής υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και παρόλα αυτά εμείς ε, καθησυχασμένοι έχουμε ζητήσει μια αύξηση 17% του Ταμείου Συνοχής. Λοιπόν, δεν είμαστε σε θέση σήμερα να συζητήσουμε προς το παρόν τα θέματα των ιδίων πόρων, της αύξησης των ιδίων πόρων ή οιεσδήποτε άλλες προτάσεις για τους ίδιους πόρους, εφόσον ταυτόχρονα δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε ε, έναν αποτελεσματικό προϋπολογισμό στον Ευρωπαίο πολίτη. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο και στον εισηγητή μας. Μία σύντομη παρέμβαση, muy brevemente λέει η πρόεδρος. Και μετά φυσικά θα απαντήσει ο κύριος Επίτροπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε. Και εξάλλου γιατί οι συναδελφοί έχουν ήδη εκφράσει ουσιαστικά όλες τις ε, σκέψεις και τις ερωτήσεις που ήθελα και εγώ να διατυπώσω και που ήταν απαραίτητες. Είναι σαφές ότι στη συζήτηση αυτή υπάρχει ένα κοινό συμφέρον από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξασφαλίσουμε ότι η οι νέοι πόροι δεν θα πρέπει να είναι μονάχα τα πλεονάσματα των προηγουμένων προϋπολογισμών. Αναρωτιέμαι πώς θα καταφέρνει η Κομισιόν σε περίοδους κρίσης να βρίσκουν πάντα πλεονάσματα του προϋπολογισμού για να καλύπτουν έκτατες καταστάσεις όπως η περίπτωση του Ίτερ. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για πραγματικά νέους πόρους και δεν είναι πρόσθετη χρηματοδότηση για τη διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών. Εδώ έχουμε μια άλλη συζήτηση η οποία πρέπει να διαμειφθεί στην Επιτροπή μας. Θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι έχουμε ήδη μια σταθμισμένη θέση που έχουμε ψηφίσει όλοι για πέντε χρόνια για τη διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών. Οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της θέσης θα έπρεπε να μας να συνοδεύεται από μια βεβαιότητα για τις δυνατότητες μεταρρύ... αναθεώρησης των δημοσιονομικών προοπτικών και ευελιξίας που αυτή τη στιγμή βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι δεδομένες. Το έγγραφο της Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών προοπτικών το έγγραφο αυτό είναι περισσότερο χρήσιμο για ένα απότερο μέλλον πέραν του 2014 από ότι για το άμεσο μέλλον. Πολύ εύκολα, πολύ καλύτερα μάλλον, αντιμετωπίζει τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε νέες δημοσιονομικές προοπτικές από ότι τη μεταρρύθμιση και την αναθεώρηση των τωρινών δημοσιονομικών προοπτικών. <clears throat> Αλλά επειδή εγώ είμαι ο εισηγητής για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές, θεωρώ ότι είναι ένα καλό έγγραφο και που δεν αποκλίνει πάρα πολύ από τις δικές μας απόψεις. Έχει πολλές σημαντικές πτυχές οι οποίες μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες για το έργο της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει το δικό της έργο και εμείς πρέπει να κάνουμε και το δικό μας έργο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν υποχρεωμένη να μας παρουσιάσει ένα έγγραφο, ένα επίσημο έγγραφο, έγγραφο σκέψης όπως θέλετε να το ονομάσετε, για το ποιε θα πρέπει να είναι οι οδηγές γραμμές των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών. Εμείς από τη δική μας πλευρά πρέπει να κάνουμε το δικό μας καθήκον. Καλό θα ήταν να συμφωνούσαν και οι δύο πτυχές αλλά είναι δύσκολο να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς να υπάρχει μια προηγούμενη επαφή και ένα feedback από τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι η ειδική η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν συμπεριέλαβε καθόλου την ε, άποψη του Κοινοβουλίου, γιατί ήταν ένα έγγραφο το οποίο δεν ε, είχε αποκαλυφθεί στις πτυχέ του παρά μόνο σήμερα. Σε πολλά σημεία συμφωνούμε. Αυτά τα οποία λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσθέμενη αξία είναι ακριβώ οι ίδιε ιδέε σχεδόν που είχε διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο έγγραφο σκέψη και στο έγγραφο εργασία που θα έχετε την επόμενη εβδομάδα από τον εισηγητή μα, από τον εισηγητή σα και για τη στρατηγική του 2020 νομίζω ότι βρισκόμαστε ακριβώ στην ίδια κατεύθυνση. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί για την πολιτική της Ευρώπης 2020, αλλά συμφωνούμε όλοι ότι στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να υπάρχει η οδηγός γραμμή της Ευρώπης του 2020. Αυτό όμως δεν καλύπτει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή τα, οι 7 ναυαρχίδες, τα 7 βασικά σχέδια καλύπτουν το 43% των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλει εκεί πέρα να συμπεριλάβει και την αγροτική πολιτική και την πολιτική συνοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το πλαίσιο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό στην πραγματικότητα, πώς θα μπορέσει να συμπεριληφθεί και η αγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχή σε αυτό το πλαίσιο. Το έγγραφο της Κομισιόν επίσης είναι αρκετά σαφέ σε σχέση με αυτά τα οποία προτείνει για την πολιτική συνοχή και την αγροτική πολιτική. Ιδίω όταν λέει ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ της στρατηγικής της Ευρώπης 2020 και της πολιτικής συνοχής. Μιλάει για κριτήρια συνεκτικότητα και συγκέντρωσης. Αναφέρει το πώς θα πρέπει η πολιτική συνοχής να τροποποιήσει τους στόχους της για να προσαρμοστεί στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παράγραφο που συνάπτεται με αυτά που συζητήσαμε σήμερα για τη βελτίωση της ποιότητας των δαπανών. Δεν ξέρω για αυτούς που έχουμε διαβάσει τώρα το κείμενο προσεκτικά, κάνει σημαντική εμβελία προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επίτροπη που θα ίσως αποτελέσουν αντικείμενο διαμάχης, γιατί με κάποιο τρόπο συνδέει την ικανότητα των κρατών μελών και των περιφερειών για να αποκτούν χρηματοδότηση στο μέλλον στην η ικανότητά τους απορρόφησης των κονδυλίων αυτών και στο επίπεδο διοικητικής διάρθρωσης και αξιοπιστίας των διοικητικών τους τομών, ώστε να κάνουν μια αποτελεσματική χρησιμοποίηση αυτών των πόρων. Αυτό είναι μια σημαντική πρόταση της Κομισιόν, η οποία πρέπει να τύχει σοβαρής Εξέταση από το έγγραφο εργασία τη Επιτροπής ΣΟΡΕ. Ούτω ή αλλω εγώ σαν πρόεδρο, σαν εισηγητή, πρέπει να πω κυρία πρόεδρο ότι το έγγραφο αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Με καθησυχάζει το γεγονο ότι οι θέσει τη Κομισιόν και του Κοινοβουλίου δεν είναι πολύ διαφορετικέ τουλάχιστον σε επίπεδο γενικών αρχών. Εμεί ω πολιτική αρχή του προϋπολογισμού έχουμε το καθήκον και το δικαίωμα να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τις γενικές αρχές αλλά σας λέω και πάλι, σαν έγγραφο είναι καλό δεκτό το έγγραφο της Κομισιόν και θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ λέει και η Πρόεδρος. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι είναι μια καλή βάση εργασίας το έγγραφο αυτό για την Επιτροπή μας, αλλά δεν θεωρώ ότι εμείς δεν δώσαμε καμία συμβολή στο έγγραφο αυτό Νομίζω ότι ο κύριος Επίτροπος δεν μας ζήτησε επίσημα να συμβάλλουμε, αλλά άκουσε πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία είπαμε. Και αντανακλώνται αυτά τα οποία έχουμε δει στο έγγραφο. Και εγώ δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένη, αλλά δεν είμαι και απόλυτα απογοητευμένη. Κύριος Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι τώρα τα πειρά θα τα χαρακτήριζα φιλικά η αλήθεια είναι ότι και στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου ίσως θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις και για τους ιδίους πόρους και για προβλήματα πιο συγκεκριμένα όπως το είτε. Δεν είναι εύκολο αυτό. Εμείς κάναμε τις προτάσεις για την διορθωτική επιστολή ακριβώς επειδή λάβαμε υπόψη μας το τι δεν δαπανήθηκε στη Γεωργία. 300 περίπου εκατομμύρια. Αυτές είναι οι εξελίξεις της δαπάνες. Το θέμα είναι αν θα τα χρησιμοποιήσουμε τα ποσά αυτά για το ίτερ. και το ίδιο θα ισχύσει και το 2011. Γνωρίζουμε σε αυτή τη φάση ότι στα πλαίσια του προγραμματισμού για τον επόμενο χρόνο πάλι θα υπάρξει ένα υπόλοιπο από τη Γεωργία. Νομίζω ότι οι εξελίξεις αυτές ε, είναι ε, θετικές και θα μπορέσουμε με ευέλικτο τρόπο, είναι χρήσιμο να μπορέσουμε με ευέλικτο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τα ποσά αυτά για την ΚΑΠ η οποία είναι, θα υπάρχει ξέρετε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι ε, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και πάρα πολλές φορές υπάρχουν παρανοήσεις. Φτάνει το 40% είναι κοινοτική προχωρημένη πολιτική, είναι πάνω από το 1% του ΑΕΠ και το θέμα είναι ότι οι διαστάσεις γύρω από αυτό το, το κεφάλαιο, οι διαστάσεις που αποκτά το συγκεκριμένο κεφάλαιο, είναι κάτι το οποίο κάνει τον κόσμο να ανησυχεί. Εν πάση περιπτώσει, συνειδητοποιώ πλήρως και το σημειώνουμε αυτό, ότι το 2009 οι άμεσες επιδοτήσεις από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό ήταν περίπου το 50% των εισοδημάτων των γεωργών. Αυτό είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ουσιαστικά το πιο σημαντικό ποσοστό το οποίο πηγαίνει προς τους γεωργούς. Το θέμα λοιπόν είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύ σοβαρό πολιτικά, πρέπει να συζητηθεί, να δούμε τι θα κάνουμε με την ύπεθρο χώρα που συρρυκνώνεται εν μέρη. Μπορεί βέβαια οι διαστάσεις να μειωθούν από το 2012, από τη σήμερα οι πιστώσεις για το κομμάτι του προϋπολογισμού που αφορά τη γεωργία και εγώ προέρχομαι από μια χώρα γεωργική εν και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν τέτοιες χώρες στην Ευρώπη ακόμα και σήμερα. Και είναι ένα πρόβλημα αυτό που θα χαρακτηρίσει τις ε, συζητήσεις στο μέλλον. Η κυρία Ζαμπάλα. τίθεται το θέμα και από πολλούς συναδέλφους πώς θα αναγνώσει κανείς ε, το συγκεκριμένο έγγραφο. Δεν μιλάμε για μία αναθεώρηση, για μία πιθανή αναθεώρηση μιλάμε, μια επανεξέταση περισσότερο. Αυτό το οποίο θα έλεγε κανείς στα πλαίσια αυτής της επανεξέτασης είναι κάποιες ρυθμίσεις για τις αρχές, να είναι συμβατές οι αλλαγές με τις αρχές του 2020 έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία, τεχνολογία, υποδομές, αηφόρος ανάπτυξη, αντιμετώπιση μετρίαση συνεπειών κλιματολογικών αλλαγών, συνοχή και καινοτομίες γενικότερα. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτές οι αρχές οι δημοσιονομικές εφαρμόζονται σύμφωνα με αυτά τα οποία περιλαμβάνει η ατζέντα για το 2020. Υπάρχει επίσης και εν μέρη μια πολύ μικρή αλλαγή για την προσαρμογή στη Λισαβόνα. Υπάρχουν και συγκεκριμένα ποσά πρακτικά, όχι μόνο προς υπόμνηση, όπως ε, η εκκίνηση λειτουργίας της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Αυτό δεν είναι θεωρητικό, αφορά πιστώσεις, αφορά τον προϋπολογισμό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μια πάρα πολύ απτή και ακριβή προσαρμογή στις καινούργιες συνθήκες. Το πώς να διαβάσει το έγγραφο αυτό. Έναρξη διαπραγματεύσεων, δυνατότητες επιλογής και όχι προκαταλήψεις. Αυτή είναι η στόχη εμείς δεν θέλουμε να προκαλέσουμε μια σαφέστατη αντίδραση από πλευράς του Συμβουλίου, μια ξεκάθαρη δήλωση για το 2011 του Συμβουλίου που θα σκοτώσει από εδώ και πέρα τη συζήτηση. Αυτό θα ήταν ε, λάθος το να προκαλέσουμε το Συμβούλιο έτσι, έτσι ώστε στο τέλος του χρόνου να υπάρξουν ε, οξύες αντιδράσεις ε, και να μην ξεκινήσει ουσιαστική συζήτηση για το 2011. Δεν το θέλουμε αυτό. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε αρκετά ισορροπημένοι, πολύ επιφυλακτικοί, βαρετοί σε σχέση με τον τρόπο που παρουσιάζουμε το έγγραφο, αλλά να ανοίξουμε κάποιες επιλογές και σκέψεις για το μέλλον. Αυτό που είπατε ότι δεν παίρνουμε μαθήματα από το παρελθόν. Όχι, νομίζω ότι τα μαθήματα από την ευελιξία σαν παράδειγμα ε, δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Έχουμε βρει αρκετά ποσά με τον τρόπο αυτό. Άνω των 80 εκατομμυρίων αν άκουσα καλά. Και είναι ένας πολύ πρακτικός τρόπος αντίδρασης αυτός και θα δείτε στο κείμενο αυτό ε, κάποια στοιχεία σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο είναι αργό μέσο, αδύναμο μέσο εσωτερικά, το οποίο θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο και εδώ τίθεται το παράδειγμα της καταστροφής στην Ουγγαρία. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε με το ταμείο αυτό για την Ουγγαρία, γιατί δεν θεωρείται φυσική καταστροφή, αλλά ανθρωπογενής φυσική καταστροφή. Με συνέπειες στο περιβάλλον. Οπότε είμαστε δεσμευμένοι, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ταμείο αυτό. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να το κινητοποιήσουμε με διαφορετικό τρόπο και να το κάνουμε και πιο ευέλικτο, όχι πιο ε, σημαντικό οικονομικά. Στον κατάλογο των ιδίων πόρων έχουμε δύο επιλογές για τον τομέα των χρηματοπιστωτικών Έχουμε τον φόρο ε, και τον φόρο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Εάν δεν υπάρξει μια συμφωνία γύρω από αυτό και ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, τότε θα υπάρξουν ε, στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό στην αγορά αυτή. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, πολλές αυξήσεις κινδύνου μετακινήσεων επιχειρήσεων, αναχωρήσεων από την Ευρώπη Συμφωνώ επίσης με κάποιες διαπιστώσεις ε, σχετικά με την αποδέσμευση του προϋπολογισμού από την παρούσα κρίση. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν αποδιοπομπαίος τράγος για τις ανεπάρκειες των φορολογικών ευρωπαϊκών συστημάτων. Δεν θα πρέπει να κατηγορηθεί ο προϋπολογισμός για τα ελλείμματα των κρατών μελών τα οποία υπάρχουν εδώ και χρόνια. Προφανώς και τα λαμβάνουμε υπόψη μας αλλά πρέπει να στρέψουμε τις ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Και έτσι θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των χρηματαγορών. Θα πρέπει απλά να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία έχουμε πει ότι θα εφαρμόσουμε. Τα συζητήσαμε και στο παρελθόν αυτό. Ευχαριστώ τον κύριο Χάγγελον για τα θετικά του σχόλια. Υπήρχε ένα λάθος στην ανακοίνωση τύπου σχετικά με τα μαθήματα του μέλλοντος όπως έλεγε ο τίτλος αλλά στην ουσία αν διαβάσετε το περιεχόμενο τα μαθήματα τα παίρνει κανείς και τα βγάζει από τη σημερινή πολιτική. Για την κυρία Τρούπελ και η σχέση με την πολιτική. Προφανώς και υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις αιτήσιες διαδικασίες, στη θέση της Ευρώπης, στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα επόμενα χρόνια, από το 2012 μέχρι το 2013 και το 2013. Η δική μου θέση είναι ότι προφανώς οι γραμμές προς υπόμνηση και δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί βέβαια στα πλαίσια της τελικής συνδιαλλαγής αλλά αυτό το οποίο είναι ο βασικός στόχος για να είμαι ειλικρινής θα είναι το Κοινοβούλιο στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων από την αρχή μέχρι το τέλος ε, και αναφέρουμε στις διαπραγματεύσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Όχι να ελέγχει απλά το Κοινοβούλιο με τα ψηφίσματά του όταν κλείσουν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος και μέσω της συνδιαλλαγής για το 2011. Εγώ δεν είμαι ουδέτερος βέβαια, είμαι προκατηλημένος εισαγωγικά σε σχέση με αυτό. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να είναι εταίρος στις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια των διακυβερνητικών επαφών, γιατί αλλιώς θα είναι καθυστερημένη η παρέμβασή του, οι αποφάσεις θα έχουν λυθεί και θα μιλάμε για τα υπόλοιπα μόνο και όχι για τα ποσά τα οποία θα διαμορφώσουν την εικόνα του μέλλοντος. Έχετε πάρα πολλή φαντασία, έχετε πάρα πολλά έμπειρα μέλη εδώ στο Κοινοβούλιο και θα μπορέσετε ε, να βρείτε τρόπους για, ε, για τον επηρεασμό των διαπραγματεύσεων από το 2011 ήδη στα πλαίσια της διαδικασίας. Αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο για το μέλλον παρά κάποια ψηφίσματα ή κάποιες δηλώσεις χωρίς ε, πρακτικές συνέπειες. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ίσως δεν είναι δουλειά μου αυτή να το λέω. Εγώ απλά εδώ τονίζω το ποια θα μπορούσε να είναι η σύνδεση των μελλοντικών διαπραγματεύσεων με το μέλλον και με τις θέσεις του Κοινοβουλίου στον καθορισμό των της οικονομίας του μέλλοντος. Ο κ. Σουμάνσκι αμφισβητεί κάποια τμήματα των πιστώσεων λέγοντας ότι εκεί όπου προκαλούνται κάποιες νέες συζητήσεις αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται τώρα στα πλαίσια της κρίσης. ακριβώς ε, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπουργοί Οικονομικών μας οδήγησαν στο να ξεκινήσουν οι συζητήσεις αυτές σχετικά με τη μείωση πιθανώς των άμεσων, των άμεσων πληρωμών. Αν μειωθούν οι άμεσες πληρωμές θα πρέπει να βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο παρέμβασης. Και αυτό μας οδήγησε στο να ξεκινήσουν νέες συζητήσεις μετά από τις δηλώσεις ορισμένων κυβερνήσεων στην Ευρώπη. Όλοι προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο να αλλάξουν τη σύνθεση με τους ιδίους πόρους και τις άμεσες πληρωμές, γιατί όλοι έχουν κάποιες εκκρεμότητες, όλοι έχουν υποσχεθεί κάποιες μειώσεις, 3%, 5%, 7% του ελλείμματος, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και δεν υπάρχει αντίφαση εδώ ανάμεσα σε προστιθέμενη αξία και στην δυνατότητα να να βοηθήσουμε τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Αυτά τα οποία παράγουν προς τη θέμενη αξία είναι οι υποδομές όπως τα ευρωπαϊκά δίκτυα, ή τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών, η διασφάλιση της προμήθειας ενέργειας, η άμεση αντίδραση σε φυσικές καταστροφές, έτσι ώστε οι χώρες να μην είναι μόνες τους στην αντίδραση σε τέτοιου είδους καταστροφές και φυσικά ε, καλό θα ήταν να λειτουργήσει άμεσα γιατί και αυτό θα παράξει προστιθέμενη αξία είναι η αρχή, η νέα υπηρεσία εξωτερική. Όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να είναι τμήμα του τρόπου με τον οποίο θα λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον κύριο Πόρτας τώρα. Θα συμφωνήσω μαζί σας με την παρατήρηση την οποία κάνατε, ότι αν μιλάμε για μια δεκαετή περίοδο θα πρέπει να έχουμε εγγυήσει για πραγματική αναθεώρηση. Οι εγγυήσει αυτές βασίζονται σε δύο πυλώνες. Πρώτον, να έχουμε αποθεματικό. Εγώ προτείνω το 5% υποχρεωτικό υπαθηματικό για την αναδιάρθρωση. Δεν μιλάμε για 1,003% ε, ε, ευελιξία το 5% είναι ένα υψηλό ποσοστό, σαν υποχρεωτικό ποσοστό, το οποίο θα μπορεί να αναδιαταχθεί, να αναδιαταχθεί και να αναθεωρήσει τον προϋπολογισμό μετά από κάποια χρόνια. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι η πολιτική, η πολιτική βούληση. Αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση για αναθεώρηση, δεν υπάρχει αναθεώρηση, οπότε δεν υπάρχει αποθεματικό. Για την κοινωνική διάσταση, αυτό αναφέρεται με κάποια ευαισθησία θα έλεγα. Το κοινωνικό ταμείο θα πρέπει να είναι πολύ πιο ορατό, πολύ πιο απτό και ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι τμήμα της πολιτικής συνοχής. Δεν θα πρέπει να διαχωριστεί το κοινωνικό ταμείο από το ταμείο συνοχής, αλλά θα πρέπει να είναι το πιο ορατό τμήμα της πολιτικής συνοχής. Για την κυρία Αντρέασεν, ως συνήθως αμφισβητεί την ποιότητα των δαπανών και την αποτελεσματικότητα των δαπανών. Βελτιώσεις υπάρχουν και στον τομέα της συνοχής και αυτό θα φανεί και από την επόμενη έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Να πω ότι για το 2010 σαν παράδειγμα μειώνουμε το πληρωμές κατά ένα δις. Το 2008 ήταν πέντε δις. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες ε, σημαντικές μειώσεις όχι όπως το 2008 βέβαια, αλλά κανένας δεν είναι τέλειος και προβλήματα υπάρχουν. Για τον Σαλβατόρ, ιδιαίτερα ευγενής ο συνήθως, έκανε κάποιες γενικές παρατηρήσεις, θετικές θα έλεγα. Έχουμε πολλές δυνατότητες να τα συζητάμε τα θέματα αυτά διμερώς και δεν θα σας απασχολήσω άλλο. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και για τα γενικότερα θετικά σας σχόλια. Αν υπάρχει κάτι θετικό, είμαστε πάντα έτοιμοι να το τονίσουμε, αλλά πάλα είμαστε και έτοιμοι να επικρίνουμε την Κομισιόν, εάν αυτό χρειάζεται. Αλλά η Κομισιόν μας άκουσε την άποψή μας και ο Ράιμερ Μπέγκε θέλει να πει κάτι πάρα πολύ εν συντομία. Ευχαριστώ για την ε, συζήτηση τον κύριο Επίτροπο. Απλώς κάτι για το χρονικό πλαίσιο, αν θα υπάρξουν από την πλευρά της Κομισιόν, μπορεί να μας πει η Κομισιόν, μας είπε ότι θα έχει νομοθετικές προτάσεις τον Ιούνιο, αλλά μήπως θα μπορούμε να έχουμε και μη νομοθετικού χαρακτήρα συνεισφορά από την ε, μεριά της Επιτροπής. Προτού απαντήσει ο Επίτροπος, δεν θα ήθελα και εγώ να τον αφήσω να φύγει από την αίθουσα. Έχετε κάποια ένδειξη να μας δώσετε. Το αργότερο τον Ιούνιο του 2011 λέει ο κύριος Επίτροπος, δεν ξέρουμε αν αυτό σημαίνει Μάιο, Ιούνιο ή κάτι άλλο. Προφανώς θα δοθούν και στο Κοινοβούλιο αυτές οι προτάσεις. Ενδεχομένως μπορεί να είναι και τον, και τον Απρίλιο. Αλλά το ερώτημα ήταν μήπως προηγουμένω θα μπορούσε να έχει κάποια ανακοίνωση μη νομοθετικού χαρακτήρα η Κομισιό να μας δώσει. Αρχές του 2011, Μάρτιο ή οτιδήποτε τέτοιο. Εμείς ούτως ή άλλως θα πρέπει να δώσουμε στο Κοινοβούλιο την πρόταση αυτή για την επόμενη περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών μαζί με τις νομοθετικές προτάσεις. Δεν μπορώ να σας πω τώρα ακριβώς πότε θα γίνει αυτό σε επίπεδο χρονικό. Θα το ελέγξω και θα επανέλθω. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλους τρεις ομιλητές εγώ τώρα. Μπέρμαν, Μπούτι Κόφερ και Αλίν Μακάρθι. Der Kommissar möchte jetzt entlassen werden. <laughs> Ο κύριος Επίτροπος ζητά να τον απελευθερώσουμε αν είναι δυνατόν. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για την παρουσία του, για την ελευσή του και του ευχόμαστε καλημέρα και επιτυχή και ε, επιτυχή συνέχεια και τόσο καλές συναντήσεις μαζί μας όπως σημαίνει στο μέλλον. Ο Τάις. Yeah. Um, thank you Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα μερικές ερωτήσεις προς τον Επίτροπο και αισθάνομαι λίγο απογοητευμένο τώρα που μιλάω και ο Επίτροπος έχει φύγει. Δύο παρατηρήσεις ωστόσο. Αν δούμε το κείμενο της Κομισιόν. Υπάρχει κίνδυνος να κινηθούμε προς το ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Όλοι βρίσκονται κάτι να παρηγορηθούν, αλλά όχι πραγματική επιλογή ανιαρό κείμενο το χαρακτηρίσει ο ίδιος ο Γιάννος Λεβαντόφσκι. Αν χρησιμοποιήσουμε τη στρατηγική 2020 ως κριτήριο για να κρίνουμε τις επιλογές του προπολογισμού υπάρχουν οι τίτλοι που χρειάζονται βαθιά μεταρρύθμιση. Και μια, ένας από τους πρώτους τίτλους είναι η ΚΑΠ. Μόνο το 18% της δαπάνης συμφωνεί με τους στόχους του 2020 για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι επιδοτήσεις ιδιαίτερα των εισοδημάτων δεν αποδίδουν ως αφρακαινοτομία, δημιουργία απασχόλησης, ε, αποδοτική χρήση των πόρων, που είναι στόχοι του 2020. Πρέπει να έχουμε το θάρρος και εδώ και η Κομισιόν να πάμε πέραν των ε, δεδομένων και εκτιμένων συμφερόντων. Ναι, ορισμένοι αγρότες έχουν κάλυψη από τις επιδοτήσεις, αλλά πολλοί αγρότες όχι. Υποχρέωσαν να καινοτομήσουν, να αλλάξουν την εκμετάλλευσή τους για να επιζήσουν στην αγορά και εξακολουθούν και το κάνουν αυτοί που παράγουν λαχανικά, φρούτα κλπ. Χρειάζομαστε μια νέα στρατηγική για τη γεωργία. Χρειαζόμαστε και αγρότες φυσικά και για τρόφιμα και για μη τρόφιμα παραγωγή για να έχουμε, για να, να έχουμε ένα υγιές μέλλον σε ένα σύγχρονο κόσμο με όχι τόσο πολύ καυτά καλοκαίρια και απερίμωση. Οι αγρότες έχουν μέλλον, αλλά είναι αυτό μια μεγάλη πρόκληση για μας. Μια κοινωνικά υπεύθυνη αναδιάρθρωση του τομέα αυτού με προσανατολισμό προς το μέλλον έξυπνη, μια έξυπνη βιώσιμη μεταρρύθμιση που να δώσει κίνητρα στους αγρότες πέραν των επιδοτήσεων με βάση τις προοπτικές του 2020. Δεύτερον, καινοτομία. Ωραία λόγια υπάρχουν για την καινοτομία στο έγγραφο της Κομισιόν, αλλά για να μπορούν και επιχειρηματίες και οι να καινοτομήσουν με κοινοτικά κονδύλια χρειαζόμαστε απλούς κανόνες, διαδικασίες και μέσα μια ένωση φιλική προς το χρήστη μετά από 60-70 χρόνια επιτέλους με απλές διαδικασίες, συναρμονισμένους κανόνες και συγχώνευση των κονδυλίων και ταμείων που έχουν τον ίδιο στόχο. Θα χρειάζεται κανείς να χτυπήσει λιγότερες πόρτες όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Τάις. Αλλά δεν είμαστε τελείως χωρίς την παρουσία της Κομισιόν. Ο Διευθυντής Λέμερ είναι παρόν και αν υπάρχουν ερωτήματα θα μπορούσε ακόμα και να μας δώσει απαντήσεις. Έχει το δικαίωμα να το πράξει αυτό. Εξάλλου ο Ράιν Μπουτικόφερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, αλλά δεν θέλω να λάβω το λόγο προσωπικά. Όχι, σαν πράσινος δεν μπορείτε να μιλήσετε έχει φύγει ο επίτροπο, οπότε δεν έχει και νόημα. Η Αλήν Μακάρτη. well, I understand, Chair, that... Μπορεί κάποιο άλλο να απαντήσει, ναι, μεν, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Είχαμε τρει βουλευτέ που κανονικά θα έπρεπε και αυτοί να υποβάλουν τι ερωτήσει του για να πάρουν απάντηση από τον Επίτροπο. Θα ήθελα στο μέλλον να μου δίνετε η δυνατότητα να μιλάω και να απαντάω ο Επίτροπο. Γιατί μιλάω εξ ονόματο των σοσιαλιστών. Δεν θα επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν. Θεωρώ ωστόσο ότι στο έγγραφο αυτό η Κομισιόν προσπαθεί να σκεφτεί το μη σκεπτεό. Πρέπει να σκεφτεί το τι δεν είναι δυνατό να σκεφτεί κανεί. Υπάρχει έλλειψη φιλοδοξία με δύο λόγια. Γιατί α πάρουμε πολιτική συνοχή. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε ένα νέο περιβάλλον με μεγάλη πίεση στι εθνικέ κυβερνήσει. Η περιοχή μου στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι μια από τι πιο φτωχέ περιοχέ, η σημερινή κυβέρνηση θα μειώσει τις δαπάνες συνοχής για τις περιφέρειες και δεν θα δώσει χρήματα για τις περιφερειακές δράσεις. Τι σημαίνει αυτό, αυτές οι φτωχές περιφέρειες που εξαρτώνται απόλυτα από την Ευρώπη για προστιθέμενη αξία, τι θα κάνουν. Πρέπει να σκεφτούμε αυτό που δεν είναι δυνατόν, το αδιανόητο κατά κάποιο τρόπο. Είχα μια πρόταση πριν από 10 χρόνια από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών στην Κομισιόν που είπε λόγω κακή απόδοση, λόγω προβλημάτων με κανόνες που ανάφερε πριν ο συνάδελφος στην περιφερειακή χρηματοδότηση. Ίσως η χρηματοδότηση να ήταν πολύ πιο μεγάλη με μια απλούστευση των κανόνων που θα επέτρεπε πιο αποδοτική χρήση των κονδυλίων και λιγότερη γραφειοκρατία. Και να μην χρειαζόμαστε να δούμε που θα διαθέσουμε κονδύλι που διδετέθηκαν στο τέλος της περίοδου. Μετά, οι έξι επιλογές της Κομισιόν. Λέει αυτές οι έξι επιλογές συμβάλλουν σε έξυπνη, ευέλικτο τρόπο ε, χρήσης κονδυλίων στο μέλλον. Αύξηση του ΦΠΑ για την Ένωση. Είναι άμεσος φόρος για τα νοικοκυριά, είναι πιο ορατός, πιο διαφανής. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει υποστήριξη γι' αυτό και επειδή είναι προοδευτικά φθήνων φόρος, πλήττει περισσότερο τους φτωχούς και δεν, φυσικά δεν είναι δημοφιλής ο νέος αυτός φόρος. Επίσης είμαι πολύ απογοητευμένη όπως και η Ισπανίδα συνάδελφος για το ότι η Κομισιόν απέρριψε πάνω κάτω την ιδέα, την ιδέα ενός φόρου στις χρηματοπιστωτικές πράξεις ενώ αναφέρεται ότι δεν φορολογείται αρκετά ο κλάδος αυτός έχει υπηρεσίες χωρίς ΦΠΑ και λέει ναι μεν είμαστε μεν ενός τέτοιου φόρου επί των πράξεων διεθνώς αλλά έχουμε ήδη τέτοιους φόρους αν δείτε τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ένα φόρο για τις ασφάλειες stamp duty το λέμε δεν στρέβλωσε την αγορά ούτε ε, έβαλε σε κίνδυνο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Κάτι πιο καινοτόμο έπρεπε να κάνει η Κομισιόν και όχι να απορρίπτει τα πάντα ευθύ εξ αρχή και να ανταποκρίνεται σε αυτό που είπε ότι εμεί το Μάρτιο ψηφίσαμε για τον φόρο αυτό στι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε και ζητάω από τον Επίτροπο να εκτελέσει αυτά τα πράγματα και όχι να πει όχι. Εμείς δουλέψαμε, ψηφίσαμε, η Κομισιόν πρέπει να δράσει. Για τα ευρωομόλογα. Καλή ιδέα. Να δούμε πώς θα λειτουργούν. Είναι ένα καλό εργαλείο για τις επενδύσεις και επειδή οι κυβερνήσει τώρα περικόπτουν τις επενδύσεις στην υποδομή, θα βοηθούσε αυτό την οικονομική ανάπτυξη στην Ένωση. Τι έχει να προτείνει για τα ευρωομόλογα η Κομισιόν. Τι συγκεκριμένε λύσεις υπάρχουν όπω είπε και ο επίτροπο, Και το πιο σημαντικό που θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο, μπορεί η Κομισιόν να απαντήσει. Έχουμε χώρε μέλη που υποστηρίζουν πολλά από τις νέες αυτές δράσεις, τις ψήφισαν για την εξωτερική δράση, για την εποπτική αρχή, για τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε στην Ένωση, πώς σκοπεύουν να προτείνουν έναν αντίστοιχο προπολογισμό. Ναι, να καταπολεμηθεί σπατάλη, η γραφειοκρατία. Αυτό όμως δεν είναι προπολογισμό για τι νέε αυτές δράσεις που είχαν την υποκρισία οι χώρε αυτέ να πούνε ναι, είμαστε υπέρ. Και τώρα ο Βρετανό Πρωθυπουργό την περασμένη εβδομάδα είπε όχι, όχι μόνο να παγώσει ο προπολογισμό, περικοπή τον προπολογισμό. Πώ θα το κάνουν αυτό. Και άλλε χώρε κάνουν το ίδιο. Η Κομισιόν μπορεί να του πιέσει να είναι πιο τίμιοι και ειλικρινεί και να μα επιτρέψουν να υπάρχει και προπολογισμό που είναι στο ύψο των περιστάσεων για φιλοδοξίε που ίδιε οι χώρε μέλη έθεσαν ω στόχο για το μέλλον τη Ένωση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, τελικά θέλω να σας πω ότι η Κομισιόν μας έχει στείλει μια διορθωτική επιστολή σε ό,τι αφορά τους τρεις φορείς για τις ε, ε, χρηματοπιστωτικές αγορές και για τις νέες ε, αρμοδιότητες που έχουν να επομιστούν και την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Αλλά για μένα αυτό το οποίο είναι, ήταν σαφές από αυτά που είπε η Αλήν, είναι ότι πρέπει να τονίσουμε το θέμα ότι ευρωπαϊκού χαρακτήρα καθήκοντα και αρμοδιότητες αυτή τη στιγμή περνάνε στα κράτη-μέλη. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά για όλα αυτά τα θέματα. Η Κομισιόν θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και πρέπει οι γενικές διευθύνσεις της γενικής της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε το δικό μας επίπεδο στο οποίο συνεργαζόμαστε, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και τι θα κάνουν και τα εθνικά κράτη και ξέρουμε ποια είναι η άποψή τους. Η στρατηγική της Λισαβόνας το 2000, για το 2010 δεν απέτυχε επειδή είχαμε λαθασμένες ιδέες, αλλά γιατί τα κράτη-μέλη σε επίπεδο εφαρμογής ουσιαστικά είχαν αντιφατικά και ακόμα και αντιπαραγωγική αντιμετώπιση. Δεν θέλουμε να έχουμε το ίδιο πράγμα και με τη στρατηγική 2020. Δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε τα κάτι μέλη δεν είναι έτοιμα να ε, δώσουν σάρκα και στην πολιτική αυτή του, της Ευρώπης του 2020 μέσω των δικών τους εθνικών πολιτικών. Δεν πρέπει λοιπόν να το λησμονήσουν αυτό τα κάτι μελη και οι αρμόδιοι υπουργοί. Αυτά ισχύουν και για την αγροτική πολιτική και για την περιφερειακή πολιτική και έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή τη δυσκολία. Δεν ξέρω πώς θα τα υπερβούμε όλα αυτά, ίσως θα πρέπει να είμαστε στο μέλλον λίγο πιο δημιουργικοί. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω από το παιχνίδι και τα κράτη-μέλη, τα οποία και αυτά πρέπει να συμμετάσχουν στην εξέβριση λύσης. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο. Κύριε Λέμε, έχετε το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Yes, uh, thank you. Um, just to assure the members... Uh, Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τα μέλη ότι παρακολουθούμε προσεκτικά όλες τις παρατηρήσεις σας, τις στέλνουμε τις παρατηρήσεις αυτές στον Επίτροπο και σε όλους τους Επιτρόπους και τίποτα δεν θα χαθεί ελπίζω. Να μου επιτρέψετε μου όμως να κάνω κάποιες διευκρινήσεις οι οποίες ίσως να σας είναι χρήσιμες. Πρώτον, παρατήρησα ότι σχετικά με τις νέους ιδίους πόρους και τον κατάλογο των επιλογών που υπάρχει, υπάρχει μια έκφραση που δημιουργεί κάποιες παρανοήσεις. Στον κατάλογο αυτό έχουμε την φορολογία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Είναι σαφές ότι αυτό είναι ένας τίτλος, ένα κεφάλαιο το οποίο περιλαμβάνει πολλές ιδέες. Μία από αυτές είναι ο φόρος των συναλλαγών και μία είναι ο φόρος των δραστηριοτήτων των χρηματοπιστωτικών. Αυτά είναι υποσυζήτηση, οπότε δεν θα πρέπει να πιστέψετε ότι ο φόρος ο προτινόμενος για τις συναλλαγές έχει τεθεί εκτός προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα είναι ανοιχτά και θα μπορέσουμε τους επόμενους δύο μήνες να δούμε τι μπορεί να γίνει με τον φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σαν μια δυνατότητα και να επανέλθουμε με μια ε, σε βάθος ανάλυση των επιλογών. Κοιτάξτε, διαδικαστικό λέει η κυρία Μακάρτιν. Γνωρίζω το τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είπε ότι θα υπάρξει ένας τέτοιος φόρος συναλλαγών, αλλά μόνο στα πλαίσια συμμετοχής ενός σφαιρικού τέτοιου είδους ε, παγκόσμιου φόρου. 20 χρόνια τον περιμένουμε αυτό το φόρο, 20 χρόνια περιμένουμε την πρότασή σας θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι η αναθεώρηση για τον προϋπολογισμό δεν κάνει καμία πρόταση γύρω από τον τομέα αυτό. Ο προϋπολογισμός και η αναθεώρηση για τον προϋπολογισμό κάνει κάποιες προτάσεις και ε, μία επιλογή, ε, μία από τις προτάσεις αυτές προς ανάλυση είναι ο φόρος για τις συναλλαγές. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε σε αυτή τη φάση. Παρατήρησα την πρότασή σας σχετικά με μια ε, χρηματοδότηση κατά 100%. Απλά αντέδρασα στην πρότασή σας, κυρία Μακάρτινγκ, ότι θα πρέπει να υπάρξει 100% χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό μας των πολιτικών συνοχής. Το έχουμε συζητήσει, έχουμε συζητήσει θέματα αποτελεσματικότητας, ελέγχου και έχουμε επίσης θέσει προσυζήτηση και το θέμα της συγχρηματοδότησης σαν χρήσιμο μέσο το οποίο δίνει την δυνατότητα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κρατημέλη να συνδυάσουν την επαγιοσύνη τους και στον τομέα τον οικονομικό. Μέχρι τώρα έχουμε δει το θέμα της συγχρηματοδότησης σαν ένα καλό μέσο ε, ορθής ε, διαχείρισης και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θα μπορέσει να γίνει αντικείμενο εξέτασης. Και κάποιες παρατηρήσεις ακόμα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Η εφαρμογή για τα θέματα της, ή μάλλον η συζήτηση για την εφαρμογή δείχνει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τα σωστά μέσα να αποφασίζονται έγκαιρα. Και γι' αυτό το χρονοδιάγραμμα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είμαστε στον ίδιο ρυθμό και λειτουργούμε με τον ίδιο ρυθμό που λειτουργούσαμε εδώ και πολλά χρόνια και είδαμε ότι στην αρχή της παρούσης δημοσιονομικής περίοδου ότι η εφαρμογή δεν ήταν πάρα πολύ εύκολη γιατί υπήρχαν καθυστερήσεις στην εναρκτήρια φάση. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από όλους που λαμβάνουν αποφάσεις στον τομέα αυτό να επιβάλλουν μια αυστηρή πειθαρχία σχετικά με το χρονισμό υιοθέτηση του πλαισίου και των 80 επιμέρους μέσων τα οποία θα πρέπει εσείς νομοθετικά να αποφασίσετε τα επόμενα δύο χρόνια. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν υιοθέτηση των μέτρων αυτών είναι κρίσιμο για την επιτυχία της εφαρμογής στο μέλλον. Και τέλος, μια παρατήρηση δεν θα πρέπει να κοιτάμε μόνο το δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και το δημοσιονομικό κανονισμό. Η συζήτηση για τον δημοσιονομικό κανονισμό ξέρετε ότι εξελίσσεται στην παρούσα φάση και καθορίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των κανόνων για την εφαρμογή του επόμενου δημοσιονομικού πακέτου. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία θα αποφασιστούν σήμερα θα επηρεάσουν το τι θα γίνει στο μέλλον. Βρισκόμαστε λοιπόν στην αρχή αλλά θα επηρεάσουμε την επιτυχία του μελλοντικού πλαισίου. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ. Η Αλήν δεν ξέρω τώρα που έχει πάει, αλλά όλη αυτή η ιστορία της φορολογίας ε, για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα ενός άλλου επιτρόπου ο οποίος ε, είναι αρμόδιος για τα θέματα αυτά. Αν θυμάμαι καλά είχε πει ότι πρέπει να κάνει μια έκθεση προς τους υπουργού ε, Οικονομικών ή για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είχε αφήσει να εννοηθεί ότι αυτός ο φόρος για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές δεν είναι το πιο πρόσφορο μέσο αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ο Ράιμερ για το θέμα των ιδίων πόρων καταρχήν πρέπει αυτό το θέμα να τεθεί στην ημερήσια διάταξη και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Και δεν θέλω να πω εγώ ότι αυτή είναι η λύση ή η άλλη λύση. Αλλά δεν μπορεί το Συμβούλιο εκ των προτέρων να μπλοκάρει μία επιλογή και να εμποδίζει την εξέβριση λύσεως σε αυτό το θέμα. Δεν έχει νόημα λοιπόν να μην υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις ανατολές για να καταλήξουμε σε κάποια λύση. Τώρα, για το θέμα του χρονοδιαγράμματος, όπως είπαμε. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα υπό ή υπό κυπριακή προεδρία. Εξαρτάται λοιπόν το να Όλα εξαρτώνται όχι μόνο από το χρονοδιάγραμμα της Κομισιόν, αλλά και από το να συμμετέχει το Κοινοβούλιο πλήρως στη διαδικασία και όχι την τελευταία στιγμή μονάχα να πληροφορείται από την ε, Επιτροπή και να λέει η Κομισιόν ότι έχει δεχτεί κάτι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και περιμένει και από το, Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνενέσει. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ε, ειλικρινή διαμεσολαβητή να είναι λίγο πιο θαραλέα στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει κάτι ακόμα. Είπατε εσεί και ορθά ότι πολλά προβλήματα δεν έχουν να κάνουν με, την αποφ... με τις αποφάσεις για την ε, ε, διαδικασία χρηματοδότησης αλλά για τα προγράμματα αυτά των 60 και 80 δισεκατομμυρίων ευρώ που χρειάστηκε να τύχουν Γενικότερη συζήτηση. Αλλά το ερώτημα είναι, θέλετε όλα αυτά τα 80 προγράμματα να εξεταστούν από την αρχή ή να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας ενδιάμεσης αναθεώρησης. Σκεφτείτε λοιπόν και το θέμα της ε, συνέχειας. Πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε με μεγαλύτερη ε, ταχύτητα ροή στα προγράμματα αυτά και μια πλήρη περάτωσή τους. Δεν μπορούμε λοιπόν τη στιγμή που έχουμε μια πολύ δύσκολη διαδικασία διαπραγμάτευσης να τα πετάξουμε όλα από το παράθυρο προγράμματα τα οποία έχουν λειτουργήσει στην πράξη και γι' αυτό σας παρακαλώ να έχετε έναν τρόπο που θα δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε θετικότερα τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας για το μέλλον. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Αυτό θα ήταν πολύ θετικό και από νομίζω όλοι μας θα μπορούσαμε να το δεχτούμε αυτό σε μια λογική αντιμετώπιση. Ο Σαλβαδόρο, απλώς μια σύσταση προς την Κομισιόν που αργά ή γρήγορα θα γίνει και πρόταση του εισηγητή της Επιτροπής αυτής. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι για το γεγονός ότι οι επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, όπως είπαμε και όλοι, θα πρέπει να προσαρμοστούν στη στρατηγική της Ευρώπης 2020. Αλλά παρόλα αυτά το κείμενο της Κομισιόν και η συζήτηση που διαμείβεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν περιλαμβάνει καμία ένδειξη για το μέχρι ποιο σημείο θα υπάρξει εθνική υλοποίηση της στρατηγικής 2020, αν θα υπάρξει υποχρεωτική συμπερίληψη αυτής της στρατηγικής στα εθνικά σχέδια για τα για τα επόμενα χρόνια. Αν δεν είναι κομμάτι των εθνικών σχεδίων και αν δεν υπάρχει μια παρακολούθηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ε, υλοποίησης της στρατηγικής αυτής στα εθνικά σχέδια, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο οι στόχοι οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτή τη στρατηγική και που θα είναι οι στόχοι των επομένων δημοσιονομικών προοπτικών να γίνουν πραγματικότητα στα κράτη-μέλη. Επομένω, μέσα στο πλαίσιο τη οικονομική ευκυβερνησία, μέσα στα πλαίσια του λεγόμενου ευρωπαϊκού εξαμήνου για την αξιολόγηση των προϋπολογισμών των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως θα έπρεπε η ανακοίνωση της Κομισιόν για τις δημοσιονομικές προοπτικές να αποσαφηνίζει πώς θα εξασφαλιστεί η υποχρεωτική συμπερίληψη της στρατηγικής Ευρώπης 2020 στα εθνικά κοινοβούλια και να διευκρινίσετε περαιτέρω και με ποιο τρόπο θα υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να επιτύχουν τους στόχους αυτούς μέσα στα εθνικά σχέδια. Αλλιώς πιστεύω θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μια ποιοτική αλλαγή και βελτίωση στην εκτέλεση των δημοσιονομικών προοπτικών στα εθνικά σχέδια. Αυτό αληθεύει και ελπίζω ότι και η Κομισιόν θα το συμπεριλάβει στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα για μένα. Εάν δεν γίνει πραγματικότητα κάτι τέτοιο, τότε η στρατηγική της Ευρώπης 2020, αν δεν αντιμετωπιστεί σαν μια ε, πραγματική προοπτική, σαν μια πραγματική προτεραιότητα από τα κράτη-μέλη, όλα τα λεφτά που θα δώσουμε εμεί, τα ελάχιστα λεφτά που θα δώσουμε, νομίζω ότι απλώ θα σπαταληθούν, δεν θα πάνε πουθενά. Πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά αυτό το θέμα η Κομισιό, κατά την άποψή μου. Δεν έχουμε άλλους ομιλητές. Ωραία. Τα σημεία 3 και 4 λοιπόν έχουν αντιμετωπιστεί. Εμείς είμαστε πολύ αποτελεσματικοί στη διαχείριση του χρόνου. Κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να το πούν αυτό. Το αρχικό σημείο 3, το... το έχουμε καλύψει. Θα πρέπει να συζητήσουμε όμως και για τις απόψεις μας για την μελλοντική στρατηγική της Ευρώπης 2020. Βλέπω να βρίσκεται σε ένα νέφος αμφιβολιών λιγάκι ο εισηγητής. Ήθελες κάτι να πεις, ε, Σαλβαδόρ, θέλεις να κάνεις μια γενικότερη επισκόπηση σε σχέση με τις ε, συνεισφορές όλων των συναδέλφων. Όχι. Ich weiß, dass es Working Document, das wird äh, υπήρξε βέβαια και είναι η ακρόαση που θα πρέπει να έχουμε προτού μας παρουσιάσεις το έγγραφο εργασία σου στην τελική του μορφή. Δεν ξέρω αν ήθελες να προσθέσεις κάτι για το έγγραφο προβληματισμού και τις απόψεις που διατύπωσαν οι συνάδελφοι υπομορφήν κατά κάποιο τρόπο σύνοψη σε σχέση με τα θέματα της Ευρώπης 2020. Αν πεις όχι, είναι όχι. Δεν είναι απαραίτητο. Εντάξει, θα το κάνουμε τότε. Αφού δεν θες, θα το κάνουμε. Κυρία Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει επικάλυψη της διαδικασίας συνδιαλλαγής για το προϋπολογισμό με την ε, επιτροπή αυτή, με τις συνεδρίες της Επιτροπής μας και αυτό σημαίνει μια αρνητική, αρνητική παρεμβολή. Υπάρχει πάντως η δυνατότητα να συμπεριληφθούν όλες οι απόψεις των συναδέλφων από την Επιτροπή Σούρα για την ε, στρατηγική 2020. Αλλά από την άλλη μεριά, από την πλευρά της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε το έγγραφο για την Budget Review όπου υπάρχει και η δική της πρόταση για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθούν οι νέες δημοσιονομικές προοπτικές με στόχο την επίτευξη της στρατηγικής 2020. Επομένως νομίζω ότι είναι κάπως πρόωρο το να ε, συζητήσουμε τώρα για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι μετά από την ε, επαφή με τον κύριο Επίτροπο και από τη στιγμή που θα έχω τις προτάσεις όλων των συναδέλφων που θα πρέπει να ενσωματώσω στην έκθεσή μου, στο έγγραφό μου και αφού με τη βοήθεια της γραμματείας συμπεριληφθούν στο εγγραφό μου όλα αυτά που είπαν τα μέλη της Επιτροπής μας και ο Επίτροπος, τότε θα μπορέσουμε να επανέλθουμε. Προς το παρόν λοιπόν δεν έχω να πω τίποτα. Έχουμε προχωρήσει λίγο περισσότερο για το έγγραφο αυτοεργασίας με τη συζήτηση που κάναμε με τον Επίτροπο. Ήταν λοιπόν μια συζήτηση που περιέλαβε και τη στρατηγική 2020 και τη συμπερίληψή της στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Επομένω, στο σημείο αυτό, κυρία Πρόεδρε, θα επαναλάβω για μια ακόμα φορά ότι δεν έχω τίποτα περισσότερο να πω. Gibt's noch Ευχαριστώ. Θέλει κάποιο άλλο να λάβει το λόγο. Όχι. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο 6 τώρα. Και θέλουμε να πούμε τώρα κάτι περισσότερο. Όχι. Απλώς σας υπενθυμίζω ότι η επόμενη μας συνάντηση είναι στις 22 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο από τις 7 έως τις 8.30. Εντάξει. Πάμε. Καλή διασκέδαση. Θα τα ξαναπούμε.